Good evening, colleagues. Um, we'll begin with point... Καλησπέρα, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 1 της της διάταξης και θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το σημείο 4 θα ξεκινήσει στις 8, όχι στις 8 παρατέταρτο. Αν έχετε λοιπόν αντιρρήσεις για την ατζέντα παστροποποίηση για να μου το πείτε. Ωραία, εγκρίνεται λοιπόν η μερική διάταξη. Έχουμε λοιπόν δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρωτού περνάσω στα θέματα της ε, ημερησίας να σας πω ότι έχουμε ε, διερμηνία και σε όλες τι γλώσσες εκτός από τα δανεικά, τα γαλλικά και τα μαλτέζικα. Ε, έχουμε λοιπόν δύο θέματα επί της ουσίας, ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιθέξης Ασύλου στο σημείο 3 και στο 4 Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΠΑ και το ζήτημα του Ασφαλού λιμένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση της δήλωσης του υποψηφίου που επιλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον διορισμό του ως νέος εκκληστικό ε, διευθυντή της ΕΑΣΟ. Ο κύριος Καρέρα επιλέχθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2016 για να επιτελέσει διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου και σύμφωνα με το άρθρο 30 ε, πριν από την ε, κονισμό για την ΕΑΣΟ, πριν από την διορισμό του, ο επιλεχθής ε, υποψήφιος θα κλείσει να κάνει μια δήλωση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσει. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Καρέρα να κάνει την εισαγωγική του παρουσίαση για 10 λεπτά κατά το όριο και μετά θα έχουν το λόγο οι συντονιστέ τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν, ε, φυσικά εφόσον το επιτρέπει και ο χρόνο. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο καταρχά στον κύριο Καρέρα. Σα καλωσορίζουμε. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members of the Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ μαζί σας. Ε, μετά την επιλογή μου από το ε, Διαχειριστικό Συμβούλιο της ε, ΕΑΣΟ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣΟ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις κεντρικές γραμμές που θέλω να προτείνω για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να συστηθώ. Είμαι Πορτογάλος υπήκος, Εργάζομαι πάνω από 30 χρόνια σε υψηλές διευθυντικές θέσεις σε όλο τον κόσμο. Έχω σχετική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνου με τον ΟΕΕ Εθνών σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αφρική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Ε, επίσης ήμουν στην αντίστοιχη θέση της Frontex ως ε, διευθύνων μιας ομάδας ε, ε, υψηλού επίπεδου και ήμασταν υπεύθυνοι για την αντίδραση στη, στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης καθώς επίσης και διευθυντικός τέλεχος σε σημαντικές επιχειρήσεις της Frontex. Έχω τελέσει ως σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα στην Ernst Young και στη Lloyd για 15 περίπου χρόνια. Ε, έχω ενημερώσει για, τις, ε, ε, για τα ενδεχόμενα σύγκρουση συμφερόντων άλλωστε. Πιστεύω ότι η προηγούμενη εμπειρία μου θα μου επιτρέψει να, κατα... να συνεισφέρω στο να περάσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη Ασύλου στην επόμενη φάση, τα επόμενα πέντε χρόνια. Να σας ενημερώσω, να προχωρήσω μάλλον ε, στα, για το σχέδιο των πέντε σημείων ε, που προτείνω ε, σε ό,τι αφορά την διαχείριση της υπηρεσίας. Δεν πρόκειται για πρόγραμμα εργασίας, ούτε πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο. Πρόκειται για, την, για το πρόγραμμά μου για τη διαχείριση υπηρεσίας, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και πού πρέπει να εστιάσουμε τη δουλειά μας. μετά τα γεγονότα του τελευταίου έτους, ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και με, τα, με το πρόγραμμα των 10 σημείων του Συμβουλίου τον Απρίλιο, η Κομισιόν ε, δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης. Και αυτή η ατζέντα, αυτό το θεματολόγιο δίνει σημαντικό ρόλο στην ε, ΕΑΣΟ. Ε, θα πρέπει να διαθέτουμε τους μηχανισμούς και την προετοιμασία που χρειάζεται για να ε, φέρουμε σε πέρα σε αυτό το έργο. Και αυτή τη στιγμή δεν τους διαθέτουμε ούτε καν το προσωπικό. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στα hot spots, και στην επανεγκατάσταση έτσι ώστε ε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Ιταλία. Αυτό άλλωστε ήταν και το βασικό μας έργο του τελευταίους μήνες και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Πιο αποτελεσματικά, πιο λειτουργικά, έτσι ώστε πραγματικά να δώσουμε τα αποτελέσματα που περιμένουν όλοι από εμά για την διαχείριση των σημείων εισόδου και των ροών των μεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές ανάγκες στην Ιταλία και την Ελλάδα, δηλαδή να εξειδικεύσουμε τη δράση μας. Στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα έχουμε ήδη αναπτύξει ε, κινητά γραφεία, σε πέντε γραφεία, έχουμε οκτώ γραφεία συνολικά σε όλη την Ελλάδα, σε πέντε μήνες. Ε, τα έχουμε εξοπλίσει με υπολογιστέ, ε, επικοινωνίες και εμπειρογνώμονες ε, εκεί ε, ενημερώνουμε ε, το τόπιο προσωπικό για, το, για ένα διαφορετικό τρόπο υποδοχής και διαχείρισης. Επίσης έχουμε δώσει, έχουμε παράσχει υπηρεσίες φαξ, διερμηνίας, κοινωνικές υπηρεσίες και ε, βοηθάμε στη, στα πρώτα στάδια της επανεγκατάστασης ε, και στον εντοπισμό του κατάλληλου προορισμού. Αυτό κάναμε τους πρώτους μήνες και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητά μου και ε, της ομάδας μου στη Μάλτα. Δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερη και τρίτη προτεραιότητα, είναι να συνεχίσουμε ε, τις δράσεις τις οποίες έχουμε ξεκινήσει ό,τι αφορά τον πίνακα ποιότητα και την κατάρτιση. Θα πρέπει να εξειδικευθούν αυτές οι υπηρεσίες μας στις ανάγκες του κάθε, του κάθε κράτους μέλους. Γιατί κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τις δικές της ανάγκες. Οι βαλτικές χώρες διαφέρουν από τις βαλκανικές χώρες. Οι μεσογειακές χώρες, ιδιαίτερα Ιταλία και Ελλάδα, χρειάζονται άλλου τύπου στήριξη. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις χώρες προέλευσης, ε, τις ασφαλείς χώρες προέλευσης, ε, τους όρους υποδοχής, ε, δημιουργία δικτύων και ανάλυση πληροφοριών για αυτά τα δίκτυα. Αυτά τα δύο θέματα είναι οι ε, δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα πρέπει να συνεχιστούν. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τη δράση μας και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές και χώρες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιχειρησιακή δράση, έχουμε ποιότητα, ανάλυση, ε, ανάλυση ποιότητας, ανάλυση πληροφοριών και τέλος, ναι, πρέπει να επιταχύνουν γιατί βέβαια ο χρόνος κυλάει, να σας πω και το εξής. Ε, όλοι σας γνωρίζετε τον αριθμό των συμπερασμάτων συνόδων κορυφής και συνεδριάσεων υψηλού επίπεδου τα οποία αναφέρονται σε θέματα μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες. Για παράδειγμα, ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου με τους ηγέτε των Δυτικών Βαλκανίων. Τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης και τα, το ε, πρόγραμμα δράση των 17 σημείων ζητούν, ζητεί από, το, από την ΕΑΣΟ να αναλάβει ε, σοβαρή δράση και το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχουμε συναντηθεί με τη Σερβία, με τη Μακεδονία, ε, έχουμε προσωπικό επιτόπου και τις βοηθάμε αυτές τις χώρες να διαχειρίζονται τις ζωές ε, στις 9 Νοεμβρίου έλαβε η χώρα η Σύνοδος Κορυφή της Βαλέτας και τα συμπεράσματά της είναι 15-20 σελίδες. Αν τα ανοίξετε στη μέση, ε, θα, εκεί σελίδα 7-8-9 υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα που αναφέρεται σε νέα καθήκοντα της υπηρεσίας υποστήριξης ασύλου της ΕΑΣΟ, στις χώρες προέλευσης, στην Αφρική και επιτόπου. Ε, μετά το πακέτο με την Τουρκία. Μα ζητήθηκε να εργαστούμε στην επανεισδοχή, στη στήριξη της Κομισιόν σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Αυτή ίσως είναι και η, ε, τρίτη ε, μας ομάδα δράσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουμε τη δράση μας. η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων μου έστειλε πολύ πρόσφατα μια επιστολή και ζητά την ΕΑΣΟ να ε, δώσει τη συνεισφορά της για το τι πρέπει να γίνει στην ε, πολιτική γειτονία. Ε, δεν έχουμε πολλή εμπειρία σε αυτό. Έχουμε ένα μικρό project το οποίο ολοκληρώνεται αυτό το μήνα. Έχουμε όμως εργαστεί για, την, ε, για χώρες όπως το Μαρόκο, η Τινησία και η Ορδανία στην οικοδόμηση ικανοτήτων και δυνατοτήτων ε, έχουμε λοιπόν κάποια εμπειρία συνεργασία και θέλουμε να τη διευρύνουμε. Έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια λοιπόν, την Τουρκία, την Αφρική και την πολιτική γειτονία. Όλα αυτά ε, αποτελούν μήνυμα εκ μέρους των θεσμικών οργάνων ότι η ΕΑΣΟ έχει και μια εξωτερική ε, ένα εξωτερικό ρόλο να παίξει στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη προφανώς και με το Διοικητικό Συμβούλιο μας βέβαια ε, και ενδεχομένως και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Πάντως σίγουρα έχουμε έναν ρόλο στην εξωτερική πολιτική αρχίζει ενωμένες από το 2016. Τέλος, μεγαλώνουμε και θα πρέπει να ε, επικοινωνούμε καλύτερα σε ό,τι αφορά το, ε, τη δράση μας. Ε, θα πρέπει να ενημερώνουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών, να συμμετέχουμε σε δίκτυα, να συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσει με όλους τους ενδιαφερόμενους ε, και, όλοι έχουν, και όλους όσοι έχουν κάποιο λόγο στο μεταναστευτικό. Αυτό θα το πάρω πολύ στα σοβαρά τα επόμενα πέντε χρόνια. Εσωτερικά επίσης θα πρέπει να μεγαλώσουμε. Χρειαζόμαστε ε, θέσεις, ε, υψηλές θέσεις ε, ε, διοικητικές, θέσεις. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και είμαι αποφασισμένος να αλλάξω την εσωτερική κουλτούρα ε, της υπηρεσίας. Με δύο λόγια και σε δέκα λεπτά αυτά είναι που προτείνω. Είναι μια, ένα στρατηγικό όραμα σε ό,τι αφορά την διαχειριστική μας προσέγγιση για την ΕΑΣΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσέξατε και είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καρέιδα. Θα δείτε ότι στην Επιτροπή μας γνωρίζουμε καλά τι είναι άσο και από το ξεκίνημα των τριμερών διαλόγων για την δημιουργία της υπηρεσίας υπήρχε ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των λεπτομεριών λειτουργίας της ε, υπηρεσίας σας και θα τύχετε της υποστήριξής μας στις μελλοντικές σας δράσεις. Οι συνάδελφοι έχουν το λόγο δύο λεπτά. Ο κ. Κοέγιο πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον ε, συμπατριώτη μου να του ευχηθώ καλή επιτυχία και να πω ότι ε, με εντυπωσίασε ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο μας ε, παρουσιάστηκε και μας παρουσίασε τα πέντε, τις πέντε άξονες δράσης του ε, για τη διαχείριση άσο τα επόμενα πέντε χρόνια. Ε, δεν είναι καινούριο διότι ήδη ήταν σε αυτή τη θέση εκτελών χρέη Από τη δημιουργία της ΙΑΣΟ ε, ε, έχει διπλασιάσει τον αριθμό του προσωπικού. Ε, μάλιστα ε, και πάλι στερεί διότι πολλά κράτη-μέλη καθυστερούν να παράσχουν το κατάλληλο προσωπικό. Πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι η ΆΣΟ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ε, τις προκλήσεις που έχει μπροστά της με το προσωπικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Και ποια πιστεύετε, ποιο πιστεύετε θα είναι η προκλήση του μέλλοντος ό,τι αφορά το προσωπικό. Φοβάμαι ότι η επιτόπου στο πεδίο στήριξη ε, που απαιτείται μπορεί να αλλάξει τη φύση της ε, υπηρεσίας. Διότι γίνεται πλέον μια σχεδόν ε, επιχειρησιακή υπηρεσία. Πιστεύετε ότι σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ΆΣΟ είναι επαρκές ή πιστεύετε ή συστήνετε στους νομοθέτες να μεταρρυθμίσουν το νομικό αυτό πλαίσιο. Ευχαριστώ. please. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να εξασφαλίσω ότι θα συμμετέχουν όσο πιο πολλοί συνάδελφοι γίνεται στη συζήτηση αυτή. Θα θέξω λοιπόν μόνο μία πτυχή. Η ΕΑΖΟ, εξ όσων καταλαβαίνω, αποτελεί μια υπηρεσία με βασικό καθήκον να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κοινού, λίγο πολύ κοινού, συστήματος για το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κτλ. Κοιτώντας λοιπόν το έργο του τελευταίου έτους, διαπιστώνουμε όλοι φαντάζομαι ότι η ΑΖΟ είναι μία από τις πιο μικρές υπηρεσίες και δεν έχει και το μεγαλύτερο δυνατό προπολογισμό. Να το πούμε έτσι εύσχημα. Και ακόμα και πέρσι ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ των κρατών μελών δεν ήταν κάτι απλό. Τώρα μιλάτε για την εξωτερική διάσταση και τον συντονισμό σε αυτό το επίπεδο παρά το γεγονός ότι συμφωνώ επί της αρχής για το ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική πτυχή, αυτή η εξωτερική διάσταση στην πολιτική ασύλου, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω άλλων τμήματων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ή μήπω χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε τεχνικό επίπεδο προς την ΕΑΖΟ για να μπορέσει να εκπληρωθεί και αυτή η εξωτερική διάσταση, πέρα από την ιστορική διάσταση. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια παραπάνω για το τι κάνετε τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσετε τώρα στα κράτη-μέλη και ποια θα μπορούσε να είναι η εξωτερική διάσταση και αν ε, φτάσετε στο σημείο που θα έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ κάποιων δράσεων, πού θα θέλετε να επικεντρωθείτε. Ευχαριστώ κυρία Ένστ. Um, Είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Θα σας δώσω το λόγο πάντως ως ε, λόγος του ότι είστε συντονιστής. Ε, τώρα ακούω τους συντονιστές πρώτα και μετά ε, ευχαριστώ την Κορνίλια. Τίμωθη, ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και τον κύριο Καρέιδα. Συμφωνώ με τον κύριο Κοέλιο απόλυτα. Η εισαγωγή του ήταν εξαιρετικά σαφής. Η δυσκολία εγκυται στο ότι έχει να αντιμετωπίσει τελείως ασαφή θέματα. Η σαφή είναι του σκοπού μπορεί να βοηθήσει, προφανώ. Δύο πράγματα ήθελα να θίξω. Ένα, Προφανώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη ε, της ε, πρώτης γραμμής ε, στα αιτήματα ασύλου υφίστανται τεράστια πίεση πόρων για να αντιμετωπίσουν τι απαιτείται από αυτούς και από το Δουμπλίνο. Θα ήθελα να μας πει λίγο περισσότερο ε, πώς με δεδομένους τους περιορισμένους πόρους μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που υφίστανται τις πιέσεις αυτές. Δεύτερον, παρότι εξετάσαμε προσεκτικά το θέμα της ε, μετεγκατάστασης, ήμουν και εισηγητή σχετικά, αν δείτε πώς γίνεται η μετεγκατάσταση, ποια κριτήρια υπάρχουν πέραν του απλού καταμερισμού στους αριθμούς, ποια κριτήρια ακολουθείς όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που χρειάζεται να μετεγκατασταθούν, μπορούμε να εξετάσουμε, να λάβουμε υπόψη τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, ε, τη συμβατότητα πολιτιστική ή άλλη για το που θα μετεγκατασταθεί κάποιος. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας σχετικά και αν είναι εφικτά αυτά ε, υπό τις συνθήκες της παρούσης Η κονίλια κονίλια Ernst. Ευχαριστώ. Καταρχάς μια ερώτηση έχω να κάνω. Κοιτώντας τον κανονισμό, γιατί είναι ΕΑΣΟ. Στο άρθρο υπαριθμών 30 για τον διορισμό του διευθυντή ορίζονται το εξή. Πριν από τον διορισμό του, οφείλει να παρουσιαστεί εδώ στην Επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει μια εντύπωση και η Επιτροπή. Κλοντ, προ εσένα αποκτήνω την ερώτηση. Περιμένω, περιμένω να βάλω τα ακουστικά σα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξή και προ τον Πρόεδρο γιατί θέλω να διασαφινιστεί αυτό για την υπόλοιπη τη δικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 30 της ΕΑΖΟ, του κανονισμού για την ΕΑΖΟ, είναι απαραίτητο πρώτο προβούμε σε διορισμό ο υποψήφιος να έλθει στην Επιτροπή για ακρόαση και μετά να συζητηθεί η δυνατότητα του διορισμού. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο τηρήθηκαν λοιπόν αυτές οι τυπικές διαδικασίες. Αυτό αφενό. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση, μάλλον μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση από την Ernst Young. Και θα ήθελα να ξέρω ποιε ήταν οι προτάσεις που συμπεριλήφθησαν στην εκτίμηση αυτή για την μεταρρύθμιση της ΕΑΖΟ, πέρα από αυτά που μας αναφέρετε εδώ. Και το πιο σημαντικό, κοιτώντας ε, την ε, εντολή της ΕΑΣΟ είναι η εφαρμογή της κοινή πολιτικής για το άσυλο. Σωστό αυτό. Αλλά πώς ε, μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, πώς θέλετε να το εξασφαλίσετε εσείς αυτό τη στιγμή που τα κράτη-μέλη σήμερα παραβιάζουν τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς ε, κανόνες και νόμους για το άσυλο και αυτό αφορά θέμα αναγνώρισης. Ουσιαστικά το δίνουν δεκάρα λοιπόν τα μελη για τα όσα ισχύουν σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, Κορνίλια. Ευχαριστώ, Πέδεψα τελείω το κατάλογο των συντονιστών και προσπαθούσα ταυτόχρονα να σα ακούσω. Σωστά θέτεις το θέμα του πώ ορίζεται ο διευθυντή ε, του ΕΑΖΟ μέχρι την άφηξη της επιστολής, να σας το διευκρινίσω, μέχρι το τέλος των ερωτήσεων, τι συμβαίνει. Οι συντονιστές αποφασίζουν τη συνέχεια που μπορεί να δοθεί μετά την ακρόαση. Έχουμε την επιλογή. Εγώ θα πρότεινα αύριο στους συντονιστές να λάβουν, να δουλέψουν πάνω στο σχέδιο της γνωμοδότησης ΛΥΜΠΕ βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού που του ΕΑΖΟ όπου υπάρχει ένα σχέδιο επιστολής από πλευράς μας με την γνωμοδότησή μας και βάσει των συζητήσεων που έγιναν σήμερα και των απαντήσεων του υποψήφιου. Αυτό λογικά γίνεται μετά τις ερωτήσεις προφανώς. Άρα είναι στην ημερήσια διάταξη αύριο το πρωί στους συντονιστές. Θα το εξηγούσα στο τέλος, αλλά τέλος πάντων το λέω και τώρα. Ανακάτεψα τον κατάλογο των συντονιστών, συνάδελφοι. Απλώς κάποιοι συντονιστές δεν αναφέρονται. Ε, αυτό που θα πω είναι ότι δεν θα μιλήσουν όλοι ακόμα και το θέλουν. Ρωτώ, πρώτα είναι οι συντονιστές. Δύο λεπτά όπως σας είπα. Ξεκινώ τώρα με την κυρία Μέτσολα που είναι η ασκούσα καθήκοντα συντονιστή. Ευχαριστώ Κολόντ και ευχαριστώ και τον κύριο Καρέιδα που ήρθε και απάντησε για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. προσβλέπω στο να σας συναντώ στη Μάλτα όσο περισσότερο γίνεται για την υπόλοιπη θητεία σας. Με την κατάσταση είναι το ερώτημά μου. Ό,τι είδαμε δείχνει ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ούτε τα hot spots εγώ ήμουν ε, ιδιαίτερα κριτική κατά του ΕΑΖΟ γιατί έβλεπα ότι υπήρχε ένας καταρχήν ρόλο του ΕΑΖΟ στην διευκόλυνση της μετακατάστασης που προκύπτει από τον κανονισμό δημιουργίας του γραφείου υποστήριξης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, εσείς και η ΕΑΖΟ θα πάρετε έναν πιο ενεργό ρόλο για να προωθήσετε την έννοια αυτή στα κράτη-μέλη. Τι χρειάζεται να γίνει για να λειτουργήσουν σωστά το συντομότερο δυνατό. Στην έκθεση που ετοίμασα με την κυρία Κιέγκε και την συνεργασία των σκιωδών εισηγητών από όλες τις πολιτικές ομάδες αναφέρουμε ότι θεωρούμε πως η Άζο πρέπει να είναι βασικός παράγοντας ε, κεδρών στον τομέα. Στο θέμα αυτό μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας ε, οπτική. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να προωθήσει τα καθήκοντα αυτά η ΆΖΟ σε σχέση με ό,τι δεν έχουν επιτευχθεί επαρκώς σωστά για να έχουμε μια πιο ουσιαστική υπηρεσία στο χώρο του ασύλου. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους σας που σέβεστε το χρόνο. Μακρύς ο κατάλογος. Θα κλείσω τώρα τον κατάλογο, ακόμα και για κάποιον που θέλει να μπει τώρα, που μπαίνει μετά από αυτή τη στιγμή επόμενος συντονιστής για τους πράσινους, κύριε Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί ήταν πολύ ανοιχτή και ειλικρινή η συζήτηση που είχαμε τον κύριο Καραϊρά. Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό και πιστεύω ότι είναι δύσκολο το έργο που έχετε να επιτελέσετε. Προσπαθείτε να διαχειριστείτε μία κρίση ασύλου με προσωρινό προσωπικό ουσιαστικά και με άτομα τα οποία έρχονται και φεύγουν από τα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν ε, είχα να σας απευθύνω μία ερώτηση θα ήταν ε, η εξής. Πώς μπορείτε να είστε αποτελεσματικός με αυτές τις συνθήκες, τις εποχές που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ. από η Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Καρέιρα για την παρουσίαση του προγράμματος και εγώ θα θέσω πολύ πρακτικές ερωτήσεις. Πρώτον, γενικά την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ένωση αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία της ΕΑΖΟ. Ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία στην πράξη αυτή της υπηρεσία. Τι μπορείτε να κάνετε περισσότερο δηλαδή σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να βελτιώσουμε την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Δεύτερον, τα hot spot, πιο συγκεκριμένα. Και εγώ έχω σοβαρές επιφυλάξεις, δεν νομίζω ότι είναι λύση ενδεχομένως να είναι τμήμα μιας λύσης της διαχείρισης των μεταναστευτικών οδών. Και εδώ ωστόσο έχω σοβαρές επιφυλάξεις. Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΑΖΟ στο hotspot. Με ποιο τρόπο η υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των διαδικασιών ταυτοποίησης και μετεγκατάστασης ε, βάση των ε, αποφάσεων για τη μετακατάσταση που υιοθετήθηκαν πριν από λίγους μήνες για την Ελλάδα και την ε, Ιταλία. Ε, δεν είναι εδώ συντονιστή του Άλντε, αλλά αν θέλει ο κ. Δεπρέ να μιλήσει ως Άλντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Καρέιλα για την σαφή παρουσίαση των στόχων και των φιλοδοξιών που έχει για το ΕΑΖΟ. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή που τέθηκε από τον κύριο Κοέλιο. Για να γίνει όλο το πρόγραμμα που μας παρουσιάσετε θα χρειαστείτε ή όχι προσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας και αποστολής της ΕΑΖΟ. Δεύτερον, τι μέσα δημοσιονομικά και σε επίπεδο προσωπικού θα χρειαστείτε τα επόμενα έτη. Εμείς έχουμε την καλή προαίρεση, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Δύο επιχειρησιακού χαρακτήρα ερωτήσει τώρα. Είπατε ότι κάνετε καταγραφή επιτόπου, αλλά στο σημείο μας σας λέει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες και να γίνουν πιο απλοποιημένες για να μην υπάρχει επικάλυψη των δράσεων με τα κράτη-μέλη. Τι θα πει αυτό επί της ουσίας και επιχειρησιακά. Ποια είναι τα προβλήματα επιτόπου ποιες καταστάσεις ε, θέλετε να θεραπεύσετε. Επίσης, έχετε ευθύνη καταγραφής, αλλά για την καλή για των hot spot, το ερώτημά μου είναι το εξή. Άπαξ και γίνει η καταγραφή. Καταγράφεται ο κόσμος. Διακρίνεται μεταξύ αυτών που κατά την άποψή σας έχουν πιθανές πιθανότητες να υπαχθούν στη διαδικασία σύλλου και άλλους που είναι άλλη κατηγορία, οικονομικοί μετανάστες θα έλεγα. Τόσο άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους τελευταίους όταν τους καταγράψετε. Τι γίνεται. Υπάρχει κάτι, υπάρχει, διαφοροποιούνται, τους αφήνουμε χήμα. Ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ούτω ώστε ο μηχανισμός να μην είναι απλώς ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός καταγραφής των εισερχομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ζράχο. Συνάδελφοι, Τώρα να επανέλθουμε στον κατάλογο. Ο κύριος Μίλλερ. Ο κύριος Μελό. Καλωσορίζω και συγχαίρω τον κύριο Καρέιρα. Ε, προφανώς επειδή είναι συμπατριώτης μου, αλλά και επειδή όμως ε, έχει τα κατάλληλα προσόντα, ε, έχει διατελέσει σε παρόμοιες θέσεις στο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο διορισμός του λαμβάνει χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο φράσεις, δύο υπουργών. Πρώτον της Αυστριακής Υπουργού, Ιωάννα Μιουκλάκεν και του Υπουργού Σουηδίας, Άντερς Γίγαμεν. που έλεγαν τα εξή. Πρώτον, αν η Ελλάδα που διαθέτει ένα από τους πιο ισχυρούς στόλους στην Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τα σύνορα της με την Τουρκία τότε είναι σαφές ότι θα αναθεωρηθούν τα όρια της Σέγγεν και θα περιοριστούν στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Υπουργός Σουηδίας είπε θα, όποιος δεν πληρεί τις υποχρεώσεις του θα ε, υποστεί ε, της, ε, περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ποια είναι η άποψή σας και πώς μπορείτε να συνεισφέρετε έτσι ώστε ο μηχανισμός μετεγκατάσταση να λειτουργήσει καλύτερα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και δεδομένων των δηλώσεων αυτών των Υπουργών. Δεύτερον, από τεχνολογική, διοικητική και ελεγκτική πλευρά, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που υπάρχουν ή πρέπει να τεθούν σε ισχύ, έτσι ώστε να γίνει διάκριση ανάμεσα στους ετούντες και τους δικαιούχους ασύλου, ποιοι είναι δηλαδή πρόσφυγες, και από την άλλη μεριά ποιοι είναι οι οικονομικοί μετανάστες και τρίτον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων τρομοκρατίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτή, αυτός ο διαχωρισμός και αν πιστεύετε ότι γίνεται αποτελεσματικά σήμερα ή αν χρειαζόμαστε άλλα μέσα, άλλες διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός με μεγαλύτερη ασφάλεια. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Καρέρα, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα και να σας συγχαρώ για την παρουσίασή σας. Παρακολουθώ το έργο της υπηρεσίας ε, πολύ στενά και χαίρομαι που βλέπω ότι η ΆΖΟ αναλαμβάνει όλο και πιο λειτουργικό ρόλο Κάποιες ερωτήσεις έχω να σας κάνω μετά τις εξελίξεις ε, των τελευταίων εβδομάδων. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη τα οποία ως τώρα ήταν αρκετά ανοιχτά για να αποδεχτούν ε, τον τεσάσυλο να υιοθετούν πλέον πιο περιοριστικές πολιτικές. Πώς ε, εκτιμάτε αυτές τις εξελίξεις και πώς μπορεί να βοηθήσει η ΙΑΖΟ. Στο πρόγραμμα λοιπόν των πέντε σημείων αναφέρεται και συμφωνώ ότι η ΕΑΣΟ θα πρέπει να συμβάλλει πιο πολύ στην εφαρμογή του συστήματος του Ευρωπαϊκού για, την, το άσυλο. Ποιος είναι ο ρόλος μας όμως σε ό,τι αφορά όλες τις ιδιαίτερες του αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τσετόσκι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Καραίρα για την εξαιρετική παρουσίαση που μας έκανα για την εξαιρετική παρουσίαση των στόχων αυτών. Πιστεύω ότι δεν είναι πολλοί υποψήφοι που μπορούν να το κάνουν αυτό με τόση σαφήνεια. Εγώ επισκέφτηκα την υπηρεσία σας πέρσι και γνωρίζω το πώς λειτουργεί, γνωρίζω ακριβώς το τι κάνει και πώς το κάνει και ποιες είναι, ε, ποια είναι τα ελλείμματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είσαστε εξίσου αποτελεσματικός όπως και ο προκάτοχός σας σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ άξιος και ικανός. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στην υπηρεσία σας, όχι μόνο α, εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς δεν έχουμε ακούσει, δεν έχει δοθεί αρκετή προβολή στην υπηρεσία σας, όχι όσο θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την χορήγηση απαλλαγής ε, προς τις υπηρεσίες, πολλοί πολλές ε, φωνές ε, κριτικής πολλοί επικριτέ θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρξει συγχώνευση τη με άλλε υπηρεσίε. Τι απάντηση λοιπόν θα δίνετε προ τι κριτικέ αυτέ, γιατί θα πρέπει η ΑΖΟ τα επόμενα 15 χρόνια να αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία και γιατί να παραμείνει και στη Μάλτα. Ευχαριστώ κυρία Γκόμε. Euh, Κύριε Καρέρα, θα ήθελα να ακούσω τι θα απαντήσετε στους προηγούμενους συναδελφούς. Ε, τι μέσα για παράδειγμα χρειάζεστε για να γίνει πιο επιχειρησιακή άσο και να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά της ε, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Μετά υπό το φως πληροφοριών που μου έφτασαν και που ελπίζω και πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσετε πολύ πρόσφατα ε, εξοπλισμός της Eurodac έφτασε στα ελληνικά hot spots. πολύ πρόσφατα. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο ε, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία να ε, γίνει ε, η καταγραφή χωρίς, αυτά τα, χωρίς αυτόν τον εξοπλισμό. Ε, όλος ο μηχανισμός μετεγκατάστασης άλλωστε λειτουργεί πολύ αργά ε, πλέον υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός Ιωροντάκου που σας είπα, πρέπει να έφτασε πολύ πρόσφατα. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί πιστεύετε ότι μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν την οδηγία 2001 περί προσωρινής προστασίας. Η Άσο θα μπορούσε να παρέμβει για παράδειγμα τη δημιουργία μια αερογέφυρας προκειμένου ε, να μετεγκαθίστανται αυτόματα ε, οι πρόσφυγες ε, και να ε, γλιτώσουμε από όλα αυτά τα κυκλώματα. Ε, επίσης είπατε ότι η περισσότερη Εξωτερική Δράση ζήτησε τη συνεισφορά σας για την πολιτική γειτονία. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται όλο και περισσότερο, οι υπουργοί παίρνουν μέτρα και με πρόχειρο τρόπο. Για παράδειγμα, ε, κατακρίνονται μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, οι οποίες βοηθούν τους μετανάστες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μας είπατε εσείς. Επίσης υπάρχουν Ευρωπαίοι Υπουργοί που προτείνουν τίνουν σε συναδέλφους τους οι αστυνομικές αρχές ή οι συνοριοφύλακες να πυροβολούν τους ε, ε μετανάστες. Ο κύριος Ράντε. Έφυγε. Η κυρία Τσενίτσι. <clears throat> Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Καρύδη για την παρουσίασή του. Πολύ ενδιαφέρουσα πρέπει να πω, διότι έδωσε και κάποιες ε, εικόνες για την διαχειριστική αντιμετώπιση του ΕΑΖΟ που καλείται να αναλάβει νέα καθήκοντα και αρκετά, με αρκετά φιλόδοξους στόχους. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω τι πόρους θέλει και στο νομικό πλαίσιο, δηλαδή τι πρέπει να αλλάξει τον κανονισμό τη, αλλά και σε ανθρώπινους πόρου. Τι μπορεί να κάνει, για να τι πρέπει να γίνει για να προσαρμοστεί. Κατόπιν μιλήσατε για πολλές ε, παραμέτρους ε, που απαιτούν ε, αλλαγή ρότας. Μιλήσατε για την διαχείριση ε, των ε, μεταναστευτικών ροών κυρίως στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μιλήσετε για την ε, ενίσχυση των δικτύων ανάλυση στην πολιτική γειτονία σε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Ρωτώ. Ε, η κρίση, η κριτική που μπορεί να αντιμετωπίσει τι κριτικές μπορεί, πώς θα αντιμετωπίζετε τυχόν κριτικές που θα προκύψουν. Μια πολύ πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Μιλήσατε όχι μόνο για το, τα hot spot και τη, και αλλά και για υποδοχή ετούντων άσυλο. Ρωτώ, προβλέπετε ή σκέφτεστε να προβλέψετε κάτι ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους οι εφημερίδες ε, σήμερα λένε ότι υπάρχουν 10.000 ε, ανήλικοι που έχουν χαθεί. 5.000 στην Ιταλία. Αυτό απαιτεί μια ειδική προσοχή. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την συνεργασία με την Frontex. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Κύριε Λόριστεν. Thank you. Uh, I suppose that... Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι το πώς θα καταστεί η εργασία όλων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών σε σχέση με τους πρόσφυγες πιο αποτελεσματική αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητα. το οποίο συζητιέται κάθε ημέρα και γι' αυτό λοιπόν η δική σας υπηρεσία καθίσταται όλο και πιο κεντρική σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για μια συνολική προσέγγιση, μιλάμε για μια κοινή πολιτική για τους πρόσφυγες, για το άσυλο. Μια κοινή πολιτική, για μια κοινή αποτελεσματική διαχείριση, γιατί είναι σαφές ότι το εφιστάμενο σύστημα, το σύστημα κατανομής, τα hot spots, όλα αυτά δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Το ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξή. Έχετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπόψη για το πώς μπορείτε να αναζητήσετε αποτελεσματικές λύσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχετε συγκεκριμένες ιδέες για να δημιουργήσετε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα από τη στιγμή της καταχώρησης μέχρι την ανακατανομή, την κατανομή, μέχρι και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στίβενς λέει ο πρόεδρος. Ζήτατε το λόγο, αλλά έκλεισα τον κατάλογο των ομιλητών πριν από λίγο. Πριν από λίγη ώρα και θα πρέπει να σεβαστώ το γεγονός αυτό γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την απάντηση του υποψήφιου διευθυντή της ΕΑΣΟ γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε και τη σχετική επιστολή για το διορισμό του αύριο. Αναγκαστικά λοιπόν θα μείνει κλειστό ο κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Σουίνμπεργκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρύρα που είστε μαζί μας σήμερα. Το βιογραφικό σας είναι πλουσιότατο, αλλά θα είναι αρκετό, δεδομένη της κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όσο και να είναι το προσωπικό σας, δεν είμαι σίγουρο, σίγουρη ότι θα μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματα. Είπατε ότι είχατε μια αντίστοιχη θέση στη Frontex. Γνωρίζετε λοιπόν τα πράγματα από πολύ κοντά. Γνωρίζετε όμως ότι η Frontex έχει ως ε, καθήκοντα κυρίως ε, ε, την διάσωση, να ζήτησε και τη διάσωση. Ε, το 85% τουλάχιστον των δραστηριοτήτων τα είναι εκεί. Εγνωρίζετε όμως και τους αριθμούς των ανθρώπων που εισέρχονται, των εισερχομένων. Είναι τεράστια αριθμοί. Είπατε ότι ανοίξατε οκτώ γραφεία ε, στην Ελλάδα. Που, τι, τι ακριβώς κάνουν ε, και πώς κατανέμουν, ε, πώς κατανέμουν τους πρόσφυγες. Ο στόχος ήταν 160.000 μετεγκαταστάσεις και το 2015 μετεγκαταστάθηκαν μόνο 300. 58.000 άτομα μπήκαν από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το Γενάρη του 2016. Οπότε τι σας αναμένει στο μέλλον. Δεν είμαι σίγουρος, σίγουρη ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα hot, spots. Οι τελευταίοι δύο μιλητές και παρακαλώ να είστε σύντομοι συνάδελφοι, ο κύριος Λεμπρετών. Είναι εδώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Καρέιρα, Κάνατε πολύ βολονταριστική παρουσίαση. Είπατε ότι θα κάνετε το ΕΑΖΟ λειτουργικό. Ε, έρχεστε ωστόσο σε ένα πλαίσιο που είναι εξαιρετικά κακό για τη δράση σας. Τα hot spot απέτυχαν, η Ελλάδα έχει πνιγεί στους μετανάστευς, ε, οι 105.000 θέσεις μετεγκατάστασης δεν εφαρμόζονται γιατί τα κράτη-μέλη δεν το θέλουν, η συμφωνία με την ε, Τουρκία είναι απάτη. Έπρεπε να δώσουμε τρία δις και ε, να απελευθερώσουμε τις θεωρήσεις για τους ε, Τούρκους πολίτες για τίποτα, γιατί δεν δεσμεύεται με τίποτα ο Ερδογάν. Ήρθε στο Στρασβούργο να μας πει πόσο κακή είναι οι Ευρωπαίοι και ο πολιτισμός τους. Το μόνο που θέλετε είναι να πετύχει η σύνοδο στη Βαλέτα που και αυτή απέτυχε. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να βοηθήσει επαρκώς την Αφρική για να περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών. Επίση το Σέγγεν διαλύεται. Προσωπικά χαίρομαι να σας πω την αλήθεια γι' αυτό. Κύριε Καρέιρα, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, πώς μπορείτε να ελπίζετε εύλογα να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του ΕΑΖΟ. Η κυρία Τσίνουν Χόκσταϊν. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση. Οι ερωτήσεις για την Frontex ε, τέθηκαν ήδη από συναδέλφους για ένα αποτελεσματικό σύστημα, καλύτερη λειτουργία των Honspot, ε, Μιλήσατε εισαγωγικά για τα θέματα αυτά. Ήθελα, κάποιος ανέφερε και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και το τεράστιο πρόβλημα που είναι η επίθεση, η δημιουργία, η μετατροπή των ε, ΜΚΟ σε εγκληματίες. Ξέρουμε ότι στα σύνορα πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν τις αφήξεις και αναχωρήσεις των ατόμων αυτών που μιλούν για ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορα. Στο κείμενο που μας παρουσιάσατε, στο σημείο 5, Υπάρχει ένα υποσημείο που λέει συνεργασία, ε, πιο δυναμική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών κτλ. Πείτε μας κάτι περισσότερα γι' αυτό. Πώς θα χρησιμοποιήσετε την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσουν το σύστημα, διότι αυτοί ξέρουν εξαιρετικά καλά την κατάσταση και έχουν μεγάλη εμπειρία και μπορεί να έχουν και ιδέες για το πώς μπορεί να γίνουν καλύτερες, ε, πιο καινοτόμες οι δουλειές και να είναι χρήσιμοι για αυτές. Ευχαριστώ όλους γιατί όλοι σεβαστήκατε το χρόνο σας. Κύριε Καρέρια, ακούσατε και υποστήριξη και προσωπική υποστήριξη. Έχετε ένα τεράστιο καθήκον σε 10-15 λεπτά να απαντήσετε σε όλες. Και υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις. Θα θέλαμε να ακούσουμε την απάντησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, ε, πολλές ε, ήταν οι ερωτήσει και καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσει προς όλες τις ερωτήσει αυτές. Θα προσπαθήσω να θυματοποιήσω κάπως. Για παράδειγμα, πολλοί μου θέσατε το ερώτημα του πώς γίνεται με τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το θέμα δεν είναι η φιλοδοξία. Είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν μπορεί να τους αφήσει και να τους αγνοήσει η ΆΖΟ. Όλα όσα ανέφερα στην εισαγωγή μου και στα πέντε σημεία. Ιδιαίτερα ο εξωτερικός ρόλος, η εξωτερική πτυχή, την οποία θέσατε κάποιοι εξημών, δεν είναι θέμα Επιλογή της ΕΑΖΟ. Όχι. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν την κατάσταση. Γιατί η προέλευση των μεταναστών είναι... Οι προελεύσεις είναι πολύ διαφορετικές. Έχουμε την, Βόρεια, την Νότια Μεσόγειο, έχουμε μετανάστες που ενδεχομένως να ζητούν καλύτερες θέσεις εργασίες, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης έχουμε την ε, Ελλάδα και την Τουρκία ως ε, πηγή με διαφορετική σύσταση αν θέλετε των μεταναστών και εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ως προς τις εθνότητες και η μεγαλύτερη μάζα είναι πραγματικά άνθρωποι που χρήζουν διεθνούς προστασία και έτσι περνούν στην Ευρώπη. Κάποιοι από εσά αναφέρατε και ρωτήσατε πώς μπορεί να ανταπεξέλθει η ΕΑΖΟ και κατά πόσο χρειαζόμαστε πιο πολλού πόρου. Ναι, χρειαζόμαστε πιο πολλού πόρου. Και αυτό φάνηκε πέρσι, στα τέλη της χρονιάς. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ ως αρμόδια επιτροπή για τις ε, πολύ θετικέ ε, τροποποιήσεις, ε, τροπολογίες που κάνατε για τη διευκόλυνση του έργου της ΕΑΖΟ στα τέλη του 2000. Έχουμε περίπου 30 νέε θέσει ε, που θα έχουν κρίσιμη σημασία για την επιτυχία τα επόμενα έτη. Αλλά δεν λάβαμε πιο πολλά χρήματα. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ε, δημιουργήθηκαν θέσει, αλλά δεν συνοδεύτηκαν από χρηματικούς πόρους. Και για πρώτη φορά λοιπόν η ΑΖΟ προετοίμασε ένα τριετέ ε, έγγραφο, το SPD, όπου θέτουμε μία προοπτική διετίας για την χώριση και την κατανομή των πόρων μας, του προσωπικού μας, των δραστηριοτήτων μας. Είναι 40 σελίδες περίπου. Στο πρώτο τμήμα εστιαζόμαστε στο 2017 και στο δεύτερο σημείο, στο δεύτερο τμήμα, ε, με πιο μακρόπρόθεσμη προοπτική, κοιτάμε τα επόμενα δύο έτη και κοιτάμε λοιπόν το πώς σχεδιάζουμε να ανταποκριθούμε στις πολλαπλές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ναι, για να έχουμε, να σας δώσουμε ένα σαφές μήνυμα. Θέλουμε να μας υποστηρίξει η Αρμόδια Επιτροπή για να έχουμε και να λάβουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να τα απεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Είτε πρόκειται για λειτουργικά καθήκοντα, για τα hot spots και ούτω καθεξή, γιατί η κρίση δεν πρόκειται να λάβει τέρμα. Και τον προηγούμενη το προηγούμενο μήνα, τον Ιανουάριο του 2016, οι ανάγκε ήταν ακόμα μεγαλύτερε από ό,τι τον Ιανουάριο του 2015. Δεν υπάρχουν ενδείξει λοιπόν ότι θα ε, μειωθεί η ροή των μεταναστών στο άμεσο μέλλον. Άρα χρειαζόμαστε πραγματικά πόρους. Ύστερα, μια δεύτερη ομάδα ερωτήσεων έχει να κάνει με πιο σοβαρά βασικά ζητήματα, όχι τόσο λειτουργικά ζητήματα κατά πόσον μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στα πλαίσια του Δουβλίνου, κατά πόσον, γιατί συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στο Δουβλίνο, κατά πόσον το τρέχον πλαίσιο μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις και απαντώ ότι ναι και αναφέρομαι στο άρθρο 5 του βασικού κανονισμού που αναφέρει ότι η ΕΑΖΟ πρέπει και έχει ευθύνη για την λειτουργική άρρωγη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα hotspots. Ήταν καινούργιο στοιχείο αυτό, αλλά το καταφέρνουμε και αυτό με περιορισμένους πόρους. Για την εντολή μας λοιπόν, για την αναθεώρηση του Δουβλίνου και για το τι κάνουμε από αυτή την άποψη. Να σας πω ότι εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στο νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Το άρθρο 5 λοιπόν μας επιτρέπει να έχουμε λειτουργική, να δίνουμε απαντήσει απαντήσεις επιτόπου και πώ το κάνουμε αυτό. Αναφέρθηκα εντάχει στο ότι αποστέλουμε προσωπικό. Έχουμε καταρτήσει δύο λειτουργικά σχέδια, ένα με την Ελλάδα και ένα με την Ιταλία για τα hot spots. Αυτό είναι λειτουργικό από τη φύση του και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητε λοιπόν, που που προγραμματίζουμε. Ένα, μια χρονική διάσταση δίνεται. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να υπογράψουμε μέχρι τον Μάρτιν του 2016 για τις δύο χώρες. Γιατί μέχρι το τέλη Ιανουαρίου έχουμε εξαρτήσει το λειτουργικό προπολογισμό για όλο το 2016 και αυτό καταδεικνύει πόσο μεγάλη έλλειψη πόρων υπάρχει. Είμαστε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Home και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη Γενική Διεύθυνση Home και θα υπάρξουν, ε, θα υπάρξουν επιπλέον πόροι. Κατά πόσον όμως θα αρκέσουν, κατά πόσον θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τον τροποποιητικό αυτό προπολογισμό δεν ξέρουμε. Αλλά πρόκειται για ένα έτος πολύ ξεχωριστό, γιατί το κατά παρελθόν δεν εργαζόμασταν, δεν λειτουργούσαμε αρκετά σωστά και δεν εξαντλούσαμε του πόρου μα. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Τι πρώτε 20 μέρε έχουμε εξοδέψει όλο τον προπολογισμό για όλο το έτος. Ναι, λοιπόν, χρειαζόμαστε πόρου. Πρέπει να αλλάξουμε άραγε το πλαίσιο και τον κανονισμό. Ίσως. Ίσως. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Όλοι συμφωνούμε και αν μπορούσα θα έβγαζα το καπέλο μου σε διευθυντής και θα σας μιλούσα με ειλικρίνεια. Τι δεν πάει καλά με το Δουβλίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχω συζητήσει με πολλούς από εσάς. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, αν θέλετε, το δικείμενο μια δεύτερη επίσκεψη. Σα παρακαλώ να με προσκαλέσετε, αν θέλετε, να συζητήσουμε και τα πολλά άλλα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Δεν λέτε το Δουβλίνο, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό να γνωρίζετε. Το... Έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε να θεωρήσει. Το τελευταίο που ακούσαμε είναι ότι θα έχουμε μία ανακοίνωση μόνο το Μάρτιο και ίσως τον Απρίλιο, ίσως και πιο μετά, θα ακολουθήσει μία πρόταση πλήρους αναθεώρησης. Όλοι ξέρουμε ότι το Δουβλίνο είχε σχεδιαστεί για μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όχι για μια κατάσταση κρίσης. Και κάποια από τα κριτήρια για την νομιμότητα, την προστασία των ατόμων, των προσφύγων, βασίζονται στις χώρες προέλευσης, στην ευθύνη της πρώτης χώρας, διέλευσης κτλ. Όλα αυτά δεν λειτουργούν στην πράξη. Κυρίως λόγω των μεγάλων ε, αριθμών ατόμων στα εξωτερικά μας σύνορα. Επειδή τα συστήματα υποδοχή σε πολλές χώρες επίσης είναι πολύ διαφορετικά, από το δικαστικό μέχρι την διεκπαιρέωση των αιτήσεων μέχρι και την, τον, τους καταλόγους χωρών προέλευσης. Και όλοι λοιπόν τα ξέρουμε αυτά. Η διάρκεια της περίοδου ε, καταχώρησης, ε, της ε, επεξεργασίας των αιτήσεων. Είναι πολλές διαφορές. Κάποιες χώρες κάνουν λίγες μέρες, κάποιες άλλες τους παίρνει παραπάνω από ένα μισή χρόνο. Έχουμε τεράστια ποσοστά αιτήσεων τα οποία δεν ε, ολοκληρώνονται. Έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο λοιπόν πλέον ε, τέτοιες αιτήσει που δεν ε, έχουν ακόμα λάβει απάντηση. Οπότε χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση του συστήματος, την υποστηρίζουμε εμείς ως ΕΑΣΟ και συμμετέχουμε στην ομάδα που εξετάζει την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Έχει συνέλθει μερικές φορές ήδη. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε. Ένα άλλο τμήμα των ερωτήσεων, η άλλη δέσμη ερωτήσεων αφορούσε το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις ροές, ιδιαίτερα μέσω της Ελλάδας. Να επαναλάβω ότι οι ομάδες μου και η Άσο γενικότερα έχουν κάνει εξαιρετικό έργο, έχουν επιδείξει εξαιρετικό παραδειγματικό έργο επιτόπου ε, και σε ό,τι αφορά ε, τον, ε, τις υπηρεσίες που προσφέρει η Άσο και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων αλλά και γενικότερα τη χρήση όλων των εργαλείων που αναπτύσσαμε τους προηγούμενους μήνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, και με πολύ επιχειρησιακό τρόπο. Αυτό ήταν ε, μεγάλη πρόκληση για μας και είμαι περήφανος που πήρα το τιμόνι πριν από μερικούς μήνες σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και δούλεψε αλλά ε, εγώ είμαι ένα γρανάζι δεν είμαι τίποτα. Ε, ε, εγώ είμαι υπέρ των πράξεων, πολύ περισσότερο από ότι υπέρ των λέξεων, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος μόνος του. Έχουμε εξαιρετικό προσωπικό και ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία πολύ αποφασιστικά μας βοηθούν και μας στέλνουν εμπειρογνώμονες. Αυτή η υποστήριξη βέβαια δεν είναι πλήρως ικανοποιητική ακόμα. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη αρρωγή. Να σας δώσω πρακτικά παραδείγματα μόνο μια μικρή πλειοψηφία των, μια μειοψηφία των κρατών μελών, κάτω από τα μισά, έχουν στείλει εμπειρογνώμονες στην ΕΑΣΟ και ακόμα και αυτά που στέλνουν το κάνουν με ένα πρόχειρο, ε, μη προγραμματισμένο τρόπο, κάτι που μας δυσκολεύει και στο δικό μας προγραμματισμό. Οπότε έχουμε κάνει έκκληση επανειλημμένως ε, στις, ε, στα κράτη-μέλη και είμαστε σε στενή επαφή με τις εθνικές υπηρεσίες ασύλου που μπορούν να μας προσφέρουν προσωπικό και νομίζω ότι κάνουμε σιγά-σιγά πρόοδο. Τώρα, σχέση με τη Frontex. Ε, έχουμε διαφορετικές εντολές η Frontex και η ASO. Το γνωρίζετε. Γνωρίζετε πολύ καλά τις διαφορές ανάμεσα σε εμά και στη Frontex. Αν έπρεπε να το συνοψίσω θα έλεγα ότι η Frontex προστατεύει τα σύνορα και εμείς προστατεύουμε τους ανθρώπους που φτάνουν μέσω των σύνορων. Διαχείριση σύνορων, διαχείριση ατόμων, ανθρώπων είναι λίγο διαφορετικές διαστάσεις. Ε, συνήθως εμείς σταματάμε στην αρχική καταγραφή, ε, μάλλον η Frontex σταματάει στην αρχική καταγραφή και από εκεί ξεκινάμε εμείς. Ενημέρωση και προστασία, αν τη δικαιούνται. Αυτό κάνουμε ξεκινάμε με ενημέρωση των ανθρώπων που φτάνουν, παράλληλα δίπλα-δίπλα με τη Frontex. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, <laughs> πολύ συγκεκριμένο όμως, με την Frontex. Ε, οι δικές μας ομάδες συνεργάστηκαν με τις ομάδες της Frontex ε, στα hotspots και ε, πέτυχε αυτό το πείραμα. Οπότε μετά την πρώτη καταγραφή και την πρώτη ενημέρωση που γίνεται από την Frontex, εκεί ξεκινάμε εμείς. Ε, εμείς ε, ενημερώνουμε τους εισερχόμενους για το πώς μπορούν να κάνουν αίτηση διεθνής προστασίας. Μετά έχουμε τη δεύτερη καταγραφή μέσω των συστημάτων της Eurodac, όπως είπε η κυρία Γκόμες. Ε, έχουμε εγκαταστήσει το software, τους υπολογιστές, τις κινητές μονάδες επικοινωνίας κλπ. Ε, και εκεί εξαντλήσαμε και τον προπολογισμό μα γι' αυτό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προπολογισμό. Θέλετε να επιταχύνω κύριε Μωράης. Καταλαβαίνω ότι σας ε, τέθησαν πολλές λεπτομερείς ερωτήσεις και μπορεί να συνεχίσετε για πολλή ώρα. Αλλά θα αναλάβω την ευθύνη και θα πω ότι θα μπορούσατε τις υπόλοιπες απαντήσεις να τις υποβάλλετε γραπτό στα μέλη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη αυτού, αυτής της πρότασης, γιατί η Επίτροπος είναι εδώ και αρκετή ώρα μαζί μας και έχουμε λιγότερο από μία ώρα στη διάθεσή μας για το επόμενο θέμα. Οπότε ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Δέκα δευτερόλεπτα μπορώ να συνεχίσω για δέκα δευτερόλεπτα. Κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες και του ανήλικους, μη συνοδευόμενου ανήλικους, του ασυνόδου ανήλικου. Και εμένα με ανησυχεί το θέμα και ένα τμήμα της ε, ε δημιουργίας ικανοτήτων ε, αφορά ακριβώς αυτές που έχουν σχέση με, τους ευάλω, με τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Ε, τεχνικές ε, εντοπισμού της προέλευσης εθνικικότητας, προ, εντοπισμός και τεχνικές ε, ε, χειρισμού των ε, ευάλωτων ομάδων κλπ. Είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να εντάξουμε στη διαδικασία ασύλου. Και συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών, γιατί είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συνεργασία. Λάμανε χώρα μία φορά το χρόνο ένα συμβουλευτικό φόρουμ στο τέλος κάθε χρονιάς. Αυτό θα αλλάξει θα δούμε πολύ πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα εμπλέκουν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το φόρουμ θα λαμβάνει χώρα τέσσερις φορές το χρόνο κάθε τρίμηνο με ένα μεγαλύτερο φόρουμ ε, στο τέλος του χρόνου γύρω στο Νοέμβριο κάθε χρονιάς. Αυτά και θα απαντήσω γραπτός για τα υπόλοιπα. Πρόεδρος. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Ένστ, που είπε στην κυρία Ένστ νωρίτερα. Αύριο το πρωί στους συντονιστές βάσει του άρθρου 30 στο 4-3-19-20 θα εξετάσουμε την ε, διαδικασία ορισμού πρότασης για, την, για τον ορισμό του κύριου Καρέιδα. Ευχαριστώ που απάντησε με λεπτομέρειες ε, ε, στις ερωτήσεις που του τέθηκαν τον κύριο Καρέιδα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ζήτησα πάρα πολλές λεπτομέρειες κάποιοι συνάδελφοι. Αν θέλει να έρθει επίτροπος για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο, ευχαριστώ ταυτόχρονα τον κύριο Καρέρα για την παρουσία του εδώ, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και το εύχομαι κάθε επιτυχία βάση του άρθρου 30 του κανονισμού ΕΑΣΟ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο. Ευχαριστώ και ελπίζω να τα πούμε. Και εγώ ευχαριστώ πρόεδρε. Καθίστε συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο για το επόμενο θέμα. Καθίστε και ξεκινήσουμε αμέσως. Colleagues, we don't have much time for this item. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι σημαντικό και γεμάτο λεπτομέρειες. Καθίστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε πάρα αυτά. Καθίστε είπα παρουσιάζεται η κατάσταση η Επίτροπος Δικαιοσύνης ε, Καταναλωτών και Ισότητας φίλων ε, την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ για την ε, συμφωνία περί ασφαλούς λιμένος μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ιδίως μετά την απόφαση ΣΕΡΜΣ. Δεν θα μιλήσω περισσότερο, ξέρω ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μας. Βέρα, έχει το λόγο. Πρόεδρε, χαίρομαι που ήρθα εδώ σήμερα για να σας ενημερώσω για τις συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ για το νέο πλαίσιο διατλαντικών ροών πληροφοριών και να ακούσω τις απόψεις για το θέμα αυτό υπόσχομαι να σας ενημερώσω υποσχέθηκα να σας ενημερώσω και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ έντονες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο ίσως να γνωρίζετε το κολέγιο θα συζητήσει την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις είπα για το θέμα αυτό και θέλω να, να σας να ενημερώσω συναδέλφους μου για το τι θα ακούσω από σας σήμερα. Η Επιτροπή είχε θέσει τον στόχο να έχει ένα ισχυρό σύστημα που θα ξεπεράσει τις αδυναμίες του παλαιού συστήματος ασφαλούς λιμένους. Οι στόχοι μας παραμένουν να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την εγγύηση των θεμελιωδών ελευθεριών όταν μεταβιβάζονται δεδομένα στη ΣΥΠΑ ή αλλού, επιτρέποντας την ροή πληροφοριών διατλαντικά ώστε να συνεχίσουν αυτά σειρές που είναι σημαντικές για την οικονομία με εχέγγυα. Το πέρυσι θέσαμε το στόχο να υλοποιηθεί σε τρεις μήνες αυτή, αυτό το πλαίσιο ε, που θα πρέπει, αυτό ήταν σαφές, να συσέβεται τους, ε, τις απαιτήσεις του ελεγκτή. Χρειαζόμαστε μια ρύθμιση βασικά διαφορετική από την, παλαιό, την παλαιά ρυθμίση για τον ασφαλή λιμένα και θα εξασφαλίσουμε την συνεχιζόμενη παρακολούθηση και αναθεώρηση των νέων ρυθμίσεων. Δεν μπορεί να είναι μια εφάπαξ απόφαση όπως αυτή που έγινε πριν από 16 χρόνια. Τους τελευταίους μήνες ε, δουλέψαμε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τους εταίρους μας από τη χώρα αυτή, ούτως ώστε να υπάρχει η δέσμευση που θα επιτρέψει την εφαρμογή μιας νέας ρυθμίσεως που θα τηρεί τις νομικές απαιτήσεις. Η αποφάση καταλληλότητας όπως ξέρετε είναι μονομερής, αλλά χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις από τη ΣΥΠΑ για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Υπογραμμίζαμε στους Αμερικανούς εταίρους ότι κάθε νέα απόφαση περί καταλληλότητας πρέπει να μπορεί να αντέξει κάποια νομική αμφισβήτηση που είναι σημαντικό και για την προστασία των δικαιωμάτων ε, του ανθρώπου αλλά και για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το κολέγιο θα συζητήσει το θέμα αύριο. Δεν είμαι λοιπόν σε θέση ακόμα να, σας, να μπω σε λεπτομέρειες για τις προτάσεις μας αλλά θα σας δώσω βασική εικόνα των ε, ζητημάτων και της κατάστασης. Οι παρατηρήσεις μου περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά θέματα για την απόφαση. Πρώτον, την ανάγκη περιορισμών και εγγυήσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση δεδομένων από τις κρατικές αρχές. Δεύτερον, ανεξάρτητη παρακολούθηση και δικαίωμα ατομικής προσφυγής στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Τρίτον, επίλυση ατομικών καταγγελιών για το πώς επιχειρήσεις επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τέταρτον ανάγκη δεσμευτικών ε, αναλήψεων υποχρεώσεων από πλευράς είπα. Για το πρώτο, εγγυήσεις και όπως ξέρετε η απόφαση ΣΡΕΠΣ κατέθεσε σαφές ότι οι υπερβάσεις αυτές θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο. Θυμίζω ότι το πλαίσιο των ήπα εξελίχθηκε μετά τις αποκαλύψεις του Σνόντεν. Υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, ε, από τον πρόεδρο Ομπάμα που έδωσε μεγαλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης και μεγαλύτερη διαφάνεια. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μας έχουμε και λαμβάνουμε γραπτές ειδικέ ε, διαβεβαιώσεις από τη ΣΥΠΑ ότι η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από κρατικέ αρχέ που όταν μεταβιβάζονται από την Ευρώπη θα περιορίζονται στο αναγκαίο και με αναλογικό τρόπο. Οι εγγυήσει, οι διαβεβαιώσει αυτέ θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρχει αδιάκριτη μαζική παρακολούθηση και ότι οι εγγυήσει ε, ε, υπέρ των ατόμων θα ισχύουν και για μη Αμερικανούς. Επιτρέψτε μου επίσης να είμαι σαφής θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και στο μέλλον. Όπως είπα στην αρχή αυτό δεν θα είναι μία απόφαση εφάπαξ αλλά το, το ξεκίνημα της παρακολούθησης. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η εμπιστοσύνη, αλλά έχουμε και καθήκον ελέγχου. Για το σκοπό αυτό θα θεσπίσουμε μια ετήσια κοινή αναθεώρηση που θα εξετάζει κάθε παράμετρο Τη συμφωνία, όπω την πρόσβαση στα δεδομένα μεταξύ και πρόσβαση στα δεδομένα από τι κρατικέ αρχέ. Επίση, θα χρησιμοποιήσουμε και άλλε διάβλου και πηγές πληροφοριών για να υπάρχει ο συνεχιζόμενο έλεγχο ατόμων, επιτεριών κοινωνία των πολιτών. Δεύτερο τομέα. Ανεξάρτητη παρακολούθηση και δικαίωμα ατομική προσφυγή. Ε, οι δυνατότητες δικαστικής προσφυγής σε ό,τι θέματα εθνικής ασφάλειας είναι περιορισμένες. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη, όπως ξέρετε. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια, ένα λειτουργικά ανεξάρτητο όργανο που θα απαντά σε καταγγελίες, ατομικές καταγγελίες Ευρω... Ευρωπαίων όταν πιστεύουν ή φοβούνται ότι οι προσωπικές τους ε, πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν παράνομα από τις ε, αρχές των ΥΠΑ στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ένα όργανο που έχει πρόσβαση σε πληροφορίες από τα εθνικά όργανα ασφάλειας. Ε, αυτό μπορεί να γίνει από έναν διαμεσολαβητή που έχει πραγματική ικανότητα δράσης και θα επιτρέπει να απαντά σε ατομικές καταγγελίες. Να στραφώ τώρα στο τρίτο θέμα, επίλυση καταγγελιών κατά επιχειρήσεων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δουλεύουμε για μια ρύθμιση που θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ατομική καταγγελία θα επιλύεται με τον α ή β τρόπο. Ιδεοδός, και όπως έδειξε και η εμπειρία, η καταγγελία θα επιλύεται από την ίδια την επιχείρηση. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που τώρα θα είναι δωρεάν. Ο πολίτης επίσης μπορεί να προσφύγει την αρχή προστασίας δεδομένων που θα παραπέμψει τις καταγγελίες στο Αμερικανικό ε, Υπουργείο Εμπορίου ή την αντίστοιχη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Μπορεί ωστόσο να υπάρχουν ανεπίλητες καταγγελίες για θέματα που δεν επιλύθηκαν από την, ε, από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή, Εμπορική Επιτροπή που εξετάζει μαζικά όχι ατομικέ καταγγελίες. Εξετάζουμε λοιπόν ένα μηχανισμό ίστατης προσέγγισης που θα επιτρέπει να επιλύονται όλες οι τελικές διαφορές μέσω ενός δεσμευτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών που επιτρέπει, που εξασφαλίζει την, ε, γιατί όπως ξέρετε το δικαίωμα στην, ε, το δικαίωμα προσφυγής ε, κατοχυρώνεται και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προφανώς στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο οι αμερικανικές αρχές προστασίας δεδομένων γιατί αυτές σέβονται τον, ε, πρέπει να σέβονται και την, ε, τον χάρτη. Οι αρχές προστασίας δεδομένων λοιπόν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν καταγγελίες είτε εμπορικού χαρακτήρα είτε εθνικής ασφάλεια, χαρακτήρα εθνικής ασφάλεια προστατεύοντας τα δικαιώματα των Ευρωπαίων όταν μεταβιβάζουν τα δεδομένα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, χρειάζεται να υπάρξουν δεσμεύσεις από τη ΣΥΠΑ που να είναι και δεσμευτικές και επίσημες αυτό δεν θα είναι διεθνή συμφωνία, αλλά μια ανταλλαγή επιστολών. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε υπογραφή στο υψηλότερο δυνατό ε, πολιτικό επίπεδο και δημοσίευση των δεσμεύσεων αυτών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το αντίστοιχο στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό θέλουμε δεσμεύσει από τη ΣΥΠΑ που θα εξασφαλίσει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία τηρεί τις απαιτήσει της ε, αποφάσεως του δικαστηρίου. Ο στόχος μας είναι, όπως είπα στο ξεκίνημα, ένα ισχυρό στέρεο σύστημα που θα επιτρέπει να επιλύεται κάθε ατομική καταγγελία, να περιορίζει την πρόσβαση των κρατικών αρχών στις πληροφορίες μόνο ότι είναι αναγκαίο και αναλογικό και η νέα αυτή ρύθμιση να παρακολουθείται σε, τακτή, σε τακτά διαστήματα με εμπλοκή των εθνικών ε, αρχών ασφαλείας και των αρχών προστασίας των δεδομένων. Δεν θα σας κρύψω ότι οι συζητήσεις δεν ήταν εύκολες. Δεν ήταν εύκολο να χτίσουμε μια στέρεη γέφυρα ανάμεσα σε δύο νομικά συστήματα με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Πιστεύω ωστόσο ότι η στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης αξίζει των προσπαθειών μας, να κάνουμε τις προσπάθειες αυτές. Και εμείς και αυτοί θα μιλήσω σήμερα το, το βράδυ αργότερα με τον Υπουργό Εμπορίου τον είπα για να συζητήσουμε τα θέματα που είναι ακόμα εκρεμή. Χρειάζεται μια περαιτέρω προσπάθεια και βασίζομαι στην υποστήριξή σας για την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τη ΣΥΠΑ το συντομότερο δυνατό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα σας ενημερώσει πλήρως για τα επόμενα βήματα κατόπιν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και Φυσικό, φυσικά θα γίνει και δήλωση από το Σώμα των Επιτρόπων αύριο. Θα υπάρχουν λοιπόν και κάποια πρόσθετα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ακόμα σήμερα. Θα περάσουμε κατευθείαν στους συντονιστές και στους συζητητές. Ε, συνάδελφοι, σας παρακαλώ να μπείτε κατευθείαν στην ουσία του θέματος και να θέσετε κατευθείαν τις ερωτήσεις σας. Δεν έχουμε χρόνο. Όλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ δύο λεπτά κατά ανώτατο όριο και αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε και ένα δεύτερο γύρο, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τις απαντήσεις της Επιτρόπου. Καταρχάς, λοιπόν, οι συντονιστές. Ο κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπό για την παρουσίασή της. Εγώ ε, ήμουν πολύ περίεργος να ακούσω το τι είχατε να πείτε για την ε, δικαστική απόφαση αυτή, την οποία δεν ήταν εύκολο να εφάρμοστε για την εθνική ασφάλεια στη ΣΥΠΑ και τα σχετικά συνταγματικά στοιχεία τα οποία θέλουμε να συμπεριληφθούν. Και νομίζω ότι ήταν σωστό το ότι δεν ακολουθήθηκαν απαραίτητα οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξανακοιτάξαμε το σύνολο του ζητήματος και αυτά που μας είπατε, ίσως όχι σε επίπεδο λεπτομέρειας, αλλά σε βάση περιπτώσει σε γενικότερο πλαίσιο, μα ικανοποιούν. Εάν εφόσον καταφέρουμε να υλοποιηθούν όλα αυτά όπως μας τα παρουσιάσατε. Νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει κάτι σημαντικό σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μετακίνηση από τη μαζική αυτή παρακολούθηση προς την στοχευμένη ε, διαβίβαση στοιχείων και δεδομένων. Αυτό θα είναι μεγάλο βήμα για να βρούμε και έτσι έναν τρόπο προκειμένου και στο θέμα της, των μυστικών υπηρεσιών να αισθάνεται μια ασφάλεια ο πολίτης και να σα ακούγονται οι ανάγκες του. Αυτό πραγματικά, αν το καταφέρετε, θα σας συγχαρώ. Εκ βάθους καρδίας, θα ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό βήμα. Για όλα αυτά που είπατε, για τους περιορισμούς τις χρήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες τη δυνατότητα ε, να εισακούεται κανείς τα θέματα επισκόπησης, όλα αυτά είναι θετικά, ακούγονται θετικά. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις λεπτομέρειες. Αλλά αν τα πετύχετε αυτά πραγματικά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ. Μπυρκίτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που μας παρουσίασε η Επίτροπος Γιούροβα ως ε, απότερο στόχο για μια νέα συμφωνία, για μια νέα διακήρυξη, δεν μπορώ παρά να το υποστηρίξω. Υποστηρίζω και τον στόχο της ασφάλισης των συνταγματικών δικαστηρίων και το να υπάρχει νομική δεθεότητα για όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχω κάποια ερωτηματικά σε θέματα λεπτομέρειας ε, και θα πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά στο τελικό κείμενο το θέμα της, του ανεξάρτητου ελέγχου, για παράδειγμα. Ποιος θα τον ε, εκτελεί και θα θέλαμε να ξέρουμε θα υπάρχει ανεξάρτητος φορέας ε, ελεγκτικός σε όλες τις ΗΠΑ, όπως το διοργανώνουμε εμείς, για παράδειγμα, στα γερμανικά κρατήδια. Θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πολιτιών, των κρατηδίων, σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια. Και στην Ευρώπη έχουμε αρκετά στοιχεία που θα έπρεπε να βελτιώσουμε. Να, βελτιώσουμε. να μην τα αναφέρουμε τώρα επιθαμένω. Πρόσβαση σε αυτά που είναι απαραίτητα. Απαραίτητα για ποιον όμως, για την βιομηχανία, την οικονομία, τις εθνικές κυβερνήσει, τις μυστικέ υπηρεσίες και ποιο τελικά θα ορίζει το τι είναι απαραίτητο ή όχι. Με ένα πολύ γενικό λόγο στόχο, καταπολέμηση της τρομοκρατίας το θέμα είναι και πώς αξιολογούμε το τι είναι απαραίτητο και ζωτική σημασία και τι όχι. Αυτό είναι πρόβλημα, θεωρώ. Ένα τελευταίο ζήτημα. Ήθελα να ρωτήσω. Πώς αξιολογείτε την τροπολογία η οποία υποβλήθηκε στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη δικαστική προσφυγή. Εγώ ερμηνεύω το κείμενο αυτό, αν και δεν έχει ακόμα εγκριθεί, ότι ουσιαστικά είμαστε αναγκασμένοι να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων. Ιδάλλως θα υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ε, στη ΣΥΠΑ. Αυτό ασφαλώς δεν συνάδει με τον γενικότερο στόχο, τον απότερο στόχο τον οποίο αναφέρατε. Ε, έχω λοιπόν πολλά μεγάλα ερωτηματικά και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά τόσο γρήγορα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει απαραίτητος να εξετάσουμε το τελικό κείμενο, γιατί νομίζω ότι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα είναι να χάσουμε τελικά στο δικαστήριο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Συνάδελφοι, ε, τους συντονιστές ε, θα ακούσουμε ε, καταρχάς. Ο κύριος Κέρκοπ δεν είναι εδώ. Η κυρία Ιντφέλτ. Uh, Να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Επιτροπό. για την ε, πολύ σκληρή δουλειά της και χαίρομαι που δεν είμαι στη θέση της. Ε, παρέλαβε αυτό το φάκελο από την προηγούμενη επιτροπή και πραγματικά είναι ένα πολύ κέριο θέμα θα έκανα δομή ότι αν είχα ξα... τι λεπτομέρειε, αλλά έχω μια-δυο πιο συγκεκριμένε και γενικότερε ερωτήσει. Ποια είναι η, ποια είναι η νομική ισχύ των δεσμεύσεων που προέρχονται από τι ΗΠΑ. Πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σα ότι δεν μιλούμε για διαπραγματεύσει, δεν μιλούμε για ένα συμβασμό, Πρόκειται για μια κατάσταση ε, στην οποία η Κομισιόν θα πρέπει να κρίνει το κατά πόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε παρέχουν επαρκή εχέγγυα, επαρκή εγγύηση. Και αναρωτιέμαι, γιατί είπατε καταρχήν ότι ε, έγιναν ήδη μεταρρυθμίσεις από τον πρόεδρο Ομπάμα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τι εγγύησει κλπ. Ποια είναι η νομική ισχύ αυτών των μεταρρυθμίσεων Έχω την εντύπωση αυτό ήταν μια μονομερής δήλωση από πλευρά του Προέδρου. Δεν ψηφίστηκε κάποιο νομοθέτημα. Μετά είπατε ότι υποβλήθηκαν γραπτές δηλώσεις και γραπτές ε, εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις από την κυβέρνηση. Αλλά σε ένα χρόνο μπορεί να έχουμε άλλη κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ο Σάντερς ή μπορεί ο Ντόναλτ Τραμπ στην εξουσία. Τι θα γίνει με αυτές. Μετά, ε, τι γίνεται με τις απαιτήσει του, της απόφασης του δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου μιλάει για περιορισμό στη συλλογή δεδομένων. Εγώ δεν βλέπω καμία, κανένα περιορισμό στη συλλογή των δεδομένων σε αυτά που είπατε. Μετά, μιλήσατε για ένα διαμεσολαβητή που θα έχει πραγματική εξουσία να ε, εξετάζει. Δηλαδή, τι, θα εξετάζει την Εθνική ε, Υπηρεσία Ασφάλειας. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Μετά μιλήσατε για υπογραφές σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο. Αν οι Αμερικάνοι είναι σοβαροί, θα πρέπει να νομοθετήσουν, αν είναι σοβαροί. Απλά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ειλικρινή και σοβαρή, γιατί αν ήταν ειλικρινή θα είχαν περάσει το νόμο περί ατομικής προσφυγής πολύ νωρίτερα, γιατί αυτός ο νόμος πραγματικά δίνει εγγύηση στους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο στους Ευρωπαίους, και στους άλλους Κατοίκου ε, κατοίκους των Πολιτείων και αλλοδαπού. Δεν νομίζω ότι είναι ειλικρινής όμως. Οπότε η Επιτροπή η Κομισιόν θα πρέπει να κρίνει όλα αυτά είναι συμβατά με την ομολογία και όχι μόνο με την, με την απόφαση της ΡΕΜΣ αλλά και με άλλε αποφάσει που ελήφθησαν αργότερα από το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μαζικές παρακολουθήσει. Όλα αυτά συμβιβάζονται με το δίκαιο, συμβιβάζονται με την νομολογία, συμβιβάζονται με τι αποφάσει και του νόμου που θα εγκρίνουμε σε λίγο. Δεν είμαι δικηγόρο. δεν μπορώ να κρίνω, δεν έχω δει τι λεπτομέρειε. αλλά ειλικρινά δεν νιώθω ήρεμη. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθεί η νομοθεσία μας. Μόνο η Κομισιόν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Και φοβάμαι ότι οποιοδήποτε ακτιβιστής, ευρωπαίος ακτιβιστής και μαζί με χιλιάδες φίλους του μπορεί να κατηγορηθεί ε, στο μέλλον ε, και όλα αυτά που είπατε δεν με καθησυχάζουν. Σα also, vielen Dank erstmal für die Darstellung. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ε, μας ε, μιλήσατε για την δικαστική απόφαση στην υπόθεση ΣΡΕΜΣ ε, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εδώ πέρα τα ξεχνάμε αυτά γρήγορα, ξέρετε. Και φροντίζετε να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε πλήρω τα θέματα αυτά. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλέ ερωτήσει που ανακύπτουν. Καταρχά, τι κάνουμε ουσιαστικά. Δεν είναι συμφωνία, δεν είναι νομοθεσία είπατε ότι πρόκειται για μία ανταλλαγή επιστολών, σημειωμάτων. Με ποιον? Είναι εντελώς αδιαφανές για μένα. Νομίζω ότι με καμία χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε μια ανταλλαγή επιστολών να αποτελέσει βάση εμπιστοσύνη για τέτοια ζητήματα, τόσο βασικά θέματα Ύστερα, για τον περιορισμό των δεδομένων, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα συμβεί αυτό το όντι. Οι συνάδελφοι από το NSA ξέρουμε ότι έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος. Ύστερα, κάθε καταγγελία θα τη χάνει επεξεργασία. Κάθε καταγγελία θα πρέπει να τη χάνει επεξεργασία από τις εταιρείε. Μήπως ανοίγουμε το κουτί τη Παντόρα, με τον τρόπο αυτό. Τι γίνεται με το νομικό πλαίσιο επίση. Μία διευκρίνηση. Και τι γίνεται με τους μη Ευρωπαίους. Συμπεριλαμβάνονται, δεν συμπεριλαμβάνονται. Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρουμε. Ειδικέ ε, γραπτέ ε, προδιαγραφέ ε, και υποσχέσει. Αυτό, τι να σα πω, είναι πάρα πολύ συνεργαστικό. Και η εμπιστοσύνη έχει τα όρια τη. Σα παρακαλώ να το Κατά δεύτερον, Ποια είναι η άποψή σας. Το Κογκρέσο λέει αν τελικά ε, βγήκε πει ότι δεν ε, προτίθεται να συμφωνήσει για τα θέματα της ε, δικαστικής προσφυγής. Τι θα γίνει με την γενικότερη συμφωνία, θα μας εκβιάσουν. Θα πούμε ναι μάλιστα, τέλεια. Επειδή είστε Αμερικανοί. Θα ήθελα να ξέρω πιο πολλές λεπτομέρειες το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. συνάδελφοι. Τώρα να ακούσουμε του δύο εισηγητέ και του υπόλοιπου ε, συναδέλφου. Να μιλήσουν όλοι, αλλά σα παρακαλώ όλοι να τηρήσετε το χρονικό όριο των δύο λεπτών. Θέλετε να πάρετε το λόγο ω συντονιστή, μάλιστα. Ως συντονίστρια. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Για να ακούσουμε και την Επιτροπή. Λόρα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, βέβαια. Οι ανησυχίες μου αφορούν καταρχάς το γεγονός ότι πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι θα γίνει η συλλογή των δεδομένων που είναι αναγκαία και σημαντικά. Τι θα πει αναγκαία και τι θα πει σημαντικά. Αφήνει πολύ χώρο ερμηνείας ε, παρακινδυνευμένης σε κάποιες περιπτώσεις. Θα έπρεπε να βάλουμε πιο δεσμευτικά πλαίσια ή έναν σαφέστερο ορισμό τι θα πει το αναγκαίο και σημαντικό για την αποφυγή κατα... καταχρήσεων. Δεύτερον, το είπαν και οι συνάδελφοι, μιλάτε για επιστολές που διαπογραφούν σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Είμαι νομικός και δύσκολο μπορώ να πιστέψω ότι μια επιστολή μπορεί να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Εφόσον δεν υπάρχει νόμος στην Αμερική, τι προστασία παρέχεται στο άτομο. Μιλάτε για προσφυγές, αλλά δεν υπάρχει νόμος. Μπορεί ένας πολίτης να υποβάλει προσφυγή βάσει μιας επιστολής. Εγώ νομικά δεν το καταλαβαίνω. Τι προστασία μπορεί να εξασφαλίζεται στα άτομα και για τους Αμερικανούς και για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Κυρία Λόριστον. Ευχαριστώ. Κλόντ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Οφείλω να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει καλά την κατάσταση. Σε, αυτό το, σε αυτή τη νέα συμφωνία, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο προστασίας είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν και ότι δεν θα χαθούν σε μια επόμενη απόφαση ΣΡΕΜΠ. Κατόπιν, δεν σχολιάσατε την διαδικασία που αφορά την τροποποίηση στη γερουσία ενός κειμένου νομικής προστασίας που λέει ότι οι πολίτες τέταρτων χωρών, τρίτων χωρών πρέπει να επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων και οι, Εθνικοί, οι Ηνωμένες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας. Αυτό είναι ένα αντεπιχείρημα, δηλαδή επιβάλλει περιορισμούς. Άρα οι δικές σας ε, προτάσεις δεν είναι πολύ πιστικές. Μπορείτε να σχολιάσετε την κατάσταση που δημιούργησε αυτή η τροπολογία. Ο Γιάννη. Ε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή που μας ενημέρωσε για τις συζητήσεις που θα μας επιτρέψουν να λάβουμε αυτή τη μονομερή αποφάση για την καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εντύπωσή μου είναι ότι πριν δούμε την ακριβή διατύπωση των διατάξεων αυτών πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχουμε μπροστά μας. Το να, λέμε, να μιλάμε για αναλογικότητα, για το δικαίωμα των μη Αμερικανών, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μη Αμερικανών πολιτών, δεν δίνει σαφή εικόνα για το τι παίζεται. Και αυτό με οδηγεί σε δύο ερωτήσεις. Πρώτον, μη Αμερικανοί πολίτες γιατί η πρόσβαση στα δεδομένα τους για λόγους εθνικής ασφάλειας θα εξετάζεται από έναν ε, διαμεσολαβητή. Πώς θα είναι αυτή η καταγγελία και ποιες θα είναι οι νομικές επιπτώσεις αυτής της καταγγελίας. Αυτό είναι σημαντικό να απαντηθεί. Ήταν μία από τη, ένα από τα βασικά επιχειρήματα του δικαστηρίου όταν αξιολόγησε το νομικό περιβάλλον στη ΣΥΠΑ ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ένδικου μέσου για πολίτες ε, μη Αμερικανούς στον τομέα αυτό. Επίσης, Μιλάτε για την εφαρμογή της συμφωνίας ε, που πάνω στο οποίο στηριζόταν ο μηχανισμός ασφαλούς λιμένα και πάνω στο οποίο θα βασίζεται και, επόμενος, ε, και επόμενη συμφωνία. Λέτε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή Εμπορίου πρέπει να εξετάζει όλες τις ε, ε όλες τις καταγγελίες Ωστόσο, μιλήσατε για, έναν, ε, για μια, ένα τελικό επίπεδο κρίσης που θα λειτουργεί με έναν τρόπο αντίστοιχο με αυτό που έχει εδώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ίστατος μηχανισμός ε, ένδικου μέσου τι θα έχει Τώρα είμαι και συγητής για τη συμφωνία Ομπρέλα. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας αυτής και του, της νομοθεσίας για, την, για τα δικαστικά ένδικα μέσα. Το ερώτημά μας είναι, τα αιτήματά μας θα, θα αντιμετωπιστούν και στη συμφωνία ομπρέλας, διότι αν αυτή η σύνδεση ισχύει θα πρέπει να ισχύει και για μας. ιδίως ό,τι αφορά την, τον περιορισμό της νομοθεσίας ε, ε, για το ένδικο μέσο σε Αμερικανούς πολίτες μόνο υπάρχει. Αν μπορεί να βρεθεί δηλαδή μια λύση για το θέμα αυτό εδώ θα έπρεπε να περάσει και στο άλλο. Κύριε Στίβενς. Ο Στίβενς. Καταρχήν ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις εξηγήσεις της. Έχω κάποιες ερωτήσεις να τις θέσω όμως. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ προέρχεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί αμοιβαιότητα και όχι μόνο καταλληλότητα. Αναμένουμε ότι τρίτες χώρες θα αντιγράψουν ε, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για όλους τους άλλους αλλοδαπούς ε, που ζουν στην ε, χώρα τους, σε ό,τι αφορά τη δικαιομαγωγή προσφυγή. προσφυγής. Θα μπορούσε επίσης η Κομισιόν να μας πει ε, τι βοήθεια προσφέρεται και τι μηχανισμοί εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια αυτή τη ενδιάμεση περίοδου, μεταβατική περίοδου. Η Κομισιόν πιστεύει ότι συμφωνία με οποιαδήποτε τρίτη χώρα θα μπορέσει να αντέξει σε δικαστική εξέταση. Τρίτον, η Επιτροπή πιστεύει ότι εδώ θα εφαρμόσουμε υψηλότερε προδιαγραφέ με τι ΗΠΑ από ό,τι εφαρμόζουμε σε άλλε συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Ευχαριστώ, κ. Bonnie. I'm Thank you very much. Thank you very much. Ευχαριστώ Επιτροπέ για τις προσπάθειές σας. Πιστεύω ότι προχωράμε, είμαι αισιόδοξο. Απ' την άλλη μεριά έχω και κάποιες αμφιβολίες. Ε, το καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε μία ευρωπαϊκή απόφαση και ένα μηχανισμό, αλλά ε, μία ε, δέσμη μηχανισμών. Επίσης είναι καλή ιδέα ε, να δημιουργήσουμε και να θεσπίσουμε τον, αυτόν τον διαμεσολαβητή, τα, τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο. Έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα ατομικής προσφυγής. Θα μπορούσατε όμως να μας περιγράψετε λίγο πιο λεπτομερώς. Δεν ξέρω αν τώρα μπορείτε να το κάνετε ή αν θα γίνει στο μέλλον. Πώς θα λειτουργήσει όμως αυτός ο μηχανισμός σχετικός με τους διαμεσολαβητές. Επίσης είναι καλή ιδέα κάθε χρόνο να ε, εξετάζεται η λειτουργία του μηχανισμού. Αλλά πώς θα γίνεται αυτή η εξέταση. Τέλος, μια αμφιβολία μου. Ε, πώς ε, εκτιμάτε, Πώς εκτιμάτε ότι είναι ειλικρινής η εκπρόσωπη των ΗΠΑ, όχι μόνο μέσω δηλώσεων, αλλά και ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Ε, τι μορφή θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις και τι ισχύει. Ο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επιτροπέ, για τις εξηγήσεις αυτές. Νομίζω ότι συγκρίνοντας την κατάσταση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από τρει μήνε, σίγουρα υπάρχουν σημαντικέ εξέλιξεις, σημαντική πρόοδο. Δεν γνωρίζουμε τι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Και θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του κατά πόσον υπάρχει συμβατότητα με το Σύνταγμα. Δεν έχει νόημα να συζητάμε τι λεπτομέρειε αν δεν έχουμε δει το συγκεκριμένο κείμενο. Ένα άλλο θέμα είναι το τι χαρακτήρα θα έχει αυτή η συμφωνία. Η ανταλλαγή απλά θα αποτελούσε ένα αρκετά στενές εργαλείο και δεν ξέρω κατά πόσον θα αρκέσει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα ανταποκρίνεται στον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ελπίζω λοιπόν να τα πετύχετε όλα αυτά. Δεν είμαι τόσο βέβαιος κατά πόσον ε, υπάρχει αυτή η επιθυμία πραγματικά από αμερικανικής πλευράς. Υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες. Αν δεν λειτουργήσει όμως αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε, έχετε κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, ένα σχέδιο β' τι σκοπεύετε να κάνετε στην περίπτωση αυτή, γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Γιώ. Λόπες Σιγκλέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ στις ευχαριστίες ε, προς την Επίτροπο για την χρησιμότητα αυτών των ε, ανταλλαγών ακόμα και για τις ε, υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις αλλά και συμφωνώ με τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν. Δύο παρατηρήσεις. Ως προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και κατόπιν την θέση σε ισχύ του νέου καθεστώτος ε, ασφαλούς ε, λιμένος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίω το ενδεχόμενο το 2000, ότι το 2016 έχει εκλογές στη ΣΥΠΑ και μιλάμε για μια ανταλλαγή επιστολών με έναν ε, πρόεδρο που τελειώνει τη θητεία του ούτως ή άλλως ε, και που δουλεύει με εχθρικές ε, πλευρές στο Κογκρέσο. Δεύτερον, μιλήσατε για την παραβίαση της συμφωνίας ε, ασφαλούς λιμένας όχι μόνο από κρατικούς φορείς, το National Security Agency, αλλά και ιδιώτες. Δηλαδή την παραβίαση κανόνων που επιβάλλονται στην Ευρώπη στις επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώς θα το δείτε αυτό με τις προοπτικές που έχουμε φέτος. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Κατανοώ τι δυσκολίε που αντιμετωπίζετε, Επιτροπέ. Είναι πραγματικά φρεχτή η κατάσταση σημερινή. Παραβιάζει το δικαίωμα μας. Και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, πρέπει να προσπαθήσετε να τα ξεπεράσετε για να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Κάτι το οποίο θα είναι νόμιμο. Αλλά ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες, όπως επισήμεναν και αρκετοί από τους αγαπητούς συναδέλφους. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω, αυτή η ιδέα του διαμεσολαβητή, θα έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει και τι γίνεται με τα κράτη-μέλη μας. Γιατί ξέρουμε ότι στα κράτη-μέλη ζητούν από τις μυστικές υπηρεσίες να κάνουν τις βρώμικες δουλειές που τους ζητούν οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αυτό μας το είπε και η υπηρεσία ΦΡΑ. Μας έχει αναφέρει σε διάφορες περιστάσεις ότι δεν υπάρχει δημοκρατικό έλεγχος σε διάφορα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η πατρίδα μου, η Πορτογαλία. Και θα θέλαμε επιτέλους κάποια, ε, κάποιο θεσμικό όργανο να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή. Γι' αυτό που είπατε τώρα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς ε, της συμφωνίας ή το κατά πόσο πρόκειτο για διεθνή συμφωνία και το καθεξής. Τα δικά μας κραμ, τη μέλη, θα το θεωρήσουν δεσμευτικό. Ακόμα και αν φέρει την υπογραφή του κύριου Γιούγκερ, του κύριου Ομπάμα, θα είναι δεσμευτικό για τα κρατη μας. Θα, ανταποκριθούν λοιπόν τα κράτη-μέλη στις ε, δεσμεύσεις τις οποίες θα αναλάβετε εσείς στη θέση τους, ο Πρόεδρος. Πριν σας δώσω το λόγο, Επίτροπε, θα ήθελα να πω το εξής. Πολλοί συνάδελφοι ε, έθεσαν το θέμα της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συμφωνίας αυτής. Δεν έχουμε ακόμα τίποτα γραπτό στα χέρια μας. Αύριο θα κάνετε την πρόταση στο Σώμα των Επιτρόπων. Συνάδελφοι, Όλοι αξιολογούμε τα όσα ακούσαμε και τα όσα υπόθηκα και δεν είναι σαφές το τι θα γίνει ακριβώς για παράδειγμα με το θέμα του διαμεσολαβητή, το πιο α, καθεστώς έχουν οι προτάσεις κτλ. Αυτό έχει επαναληφθεί. Δεν ήταν κανείς άλλος στον κατάλογο των ομιλητών. Δεν θα ακούσουμε λοιπόν κανέναν άλλο συνάδελφο. Αλλά να πω το εξή. Δεν είσαι στο κατάλογο. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγη κατανόηση και θα σας συμπεριλάβω στον επόμενο γύρο. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Δύο προτάσεις λοιπόν έχω να κάνω για να βοηθήσουμε και την Επιτροπή στο έργο της αλλά και τους εαυτούς μας να γίνει μια ειδική αχρόαση με τους ανώτατους ε, αξιωματούχους των ΙΠΑ προκειμένου με ανοιχτό χαρακτήρα και με διαφάνεια να έρθουν να μας μιλήσουν για τον διαμεσολαβητή, για παράδειγμα, κατά πόσον θα βοηθάει τον κόσμο σε ό,τι αφορά θέματα το, ατομικής προσφυγής και να υπάρξει και ένα ψήφισμα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα πολιτικό έναυσμα από πλευρά μα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι περίεργη η διαδικασία αυτή, δεν είναι διεθνή συμφωνία Είναι υβριδικού τύπου η συμφωνία αυτή θα έλεγα. Αυτό λοιπόν θα προτείνω αύριο στους συντονιστές. Για να απαντήσω στην ανησυχία που άκουσα. Επίτροπε, αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Είναι να μένω το μικρόφωνο μου. Ωραία. Ήταν αναμενόμενο η περιγραφή μου να σας φανεί ανεπαρκής. Το είπα όμως ε, από την αρχή της τοποθετησής μου ότι θα πρέπει να είμαι λίγο γενικόλογη. Κάποιοι είπατε ότι είστε δικηγόροι και οι δικηγόροι πάντοτε θέλουν να έχουν μπροστά τους το κείμενο γιατί ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Οπότε σας ζητώ ξανά συγγνώμη, λυπάμαι που σας δίνω μόνο γενικές πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας περισσότερες λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω ό,τι μπορώ να απαντήσω. Με ρωτήσατε αν εμπιστεύομαι τους συνομιλητές μου, τους ομολόγους μου. Πρέπει να τους εμπιστευτώ. Ταυτόχρονα όμως πάντοτε λέω ας ελέγχουμε κιόλας. Και αυτό που προσπαθήσαμε ήταν στη, στον τομέα του περιορισμού της ε, πρόσβασης στα δεδομένα από πλευρά των υπηρεσιών ε, εθνικής ασφάλειας απαιτήσαμε λεπτομερή περιγραφή των περιορισμών πώς προκύπτουν από την εθνική τους νομοθεσία πώς προκύπτουν από την από το προεδρικό διάγραμμα ε, ε, διάταγμα 28 ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαιρέσει με βάση οποίε οποίες υπάρχει πρόσβαση από πλευρά τη Εθνική Υπηρεσία Ασφάλεια και μα δώσανε μια πολύ λεπτομερή περιγραφή αυτών των περιορισμών. Και ξέρουμε τι, πώς κατανοούν τον όρο αναγκαίο και αναλογικό. αυτή είναι όροι δικοί μας και πρέπει να αντιληφθούμε πώς τους καταλαβαίνουν οι συνομιλητές μας. Οπότε έχουμε αυτή την περιγραφή στα χέρια μας. Είναι μια πολύ αναλυτική περιγραφή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στοχευμένη και εξειδικευμένη ε, πρόσβαση η οποία θα ε, έχει προτεραιότητα έναντι της γενικής και μαζικής πρόσβασης θα γίνεται κατ' εξαίρεση. Πρώτον, αν η εξειδικευμένη και στοχευμένη δεν είναι δυνατόν να γίνει ή αν εντοπιστεί συγκεκριμένη τάση που δεν μπορεί να ανοιχνευτεί, να εξεταστεί με στοχευμένη πρόσβαση. Πάντως η στοχευμένη πρόσβαση θα είναι ο κανόνας και η προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν ε, να ε, ε, παίξει ένα δευτερεύοντα ρόλο εναντί της μαζικής και γενικευμένης πρόσβασης. Αυτή η περιγραφή είναι ένα πράγμα όμως. Το άλλο είναι το πώς θα μπορούμε να ελέγξουμε την εφαρμογή όλων αυτών. Και γι' αυτό είπα πολύ ειλικρινά στην αρχή, η Κομισιόν έχει υποσχεθεί και δεσμεύεται να, να κάνει συνεχούς ελέγχους. Πρώτον μέσω μιας ετήσιας έκθεσης και οι εθνικοί φορείς ασφαλείας θα συνεισφέρουν σε αυτήν την έκθεση. Δεύτερον, θα ελέγχουμε μέσω των εταιριών των αριθμών των ετοιμάτων στα οποία χρειάστηκε να απαντήσουν. Θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα κανάλια ε, αναφορές από τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης, ε, εκθέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. Για μένα αυτό είναι το πιο καθόδε ζήτημα, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό ότι είναι μυστικές και δεν είναι δυνατόν να μας ενημερώνουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις έτσι ώστε να διαπιστώνουμε αν το κριτήριο της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας εφαρμόστηκε σωστά. Γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε τον διαμεσολαβητή ή την διαμεσολαβήτρια που κατόπιν αιτήματός μας θα βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της αμερικανικής ε, διοίκησης. Και ο διαμεσολαβητής αυτός ε, πρέπει, όπως ζητούμε, να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος και να έχει την εξουσία να ζητά από, τους, από τα όργανα ασφαλείας των ΗΠΑ πληροφορίε για συγκεκριμένε υποθέσεις. Εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ γιατί η μορφή του διαμεσολαβητή μας προτάθηκε ως εναλλακτική λύση πολύ πρόσφατα. Οπότε θα πρέπει να επεξεργαστούμε ακόμα τις λεπτομέρειες. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι αν υιοθετηθεί η λύση του διαμεσολαβητή, επιμένουμε ο διαμεσολαβητής να έχει πλήρεις αρμοδιότητες και ισχυρές εξουσίες να επεξεργάζεται και να απαντά στις καταγγελίες των προσώπων που θα προσφέρουν σε αυτόν και ότι θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να διαπιστώσει αν τα δεδομένα των συγκεκριμένων ατόμων δεν έτυχαν επαρκούς προστασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ασφαλή λιμένα, ε, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, οπότε δεν θα σχολιάσω γι' αυτό, αλλά είναι σαφές και από την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και από προηγούμενα πορίσματά μας, ε, είναι φανερό πως χρειάζεται μια καινούρια διευθέτηση. Έτσι θα την ονομάσουμε, όχι νέος ασφαλής λιμένας, θα την ονομάσουμε νέα διευθέτηση. Η απόφαση του, Ευρωπαϊκού, του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας βοηθάει βέβαια γιατί μας θέτει τον πύχη. Το χρειαζόμαστε μία, όμως μια καινούρια διευθέτηση γιατί είναι τεράστιος ο όγκος δεδομένων από, τις Ευρω... από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές επιχειρήσεις εμπλέκονται σε αυτές τις ροές. Με ρωτήσατε αν κάνουμε το ίδιο και σε ό,τι αφορά άλλες τρίτες χώρες. Ασφαλώς. Όταν είναι να λάβουμε μια απόφαση καταλληλότητας για μια τρίτη χώρα, εξετάζουμε αν εκεί υφίσταται ισοδύναμη ή αντίστοιχη ανάλογη προστασία με αυτήν που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζητούμε όμως οι πολιτείες να λάβουν ισχυρές νομικές δεσμεύσεις για το ότι στην Αμερικανική επικράτεια θα θεσπιστεί ένα σύστημα επαρκούς προστασίας, επαρκών εγγύσεων, έτσι ώστε να αξιολογηθεί ως ισοδύναμο αυτό σαφώς και ρητά απαιτεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μας. Δεν αναζητούμε ταυτόσιμη ίδια προστασία. Γιατί, γιατί είναι δύο διαφορετικά συστήματα που προσπαθούμε να τα ε, συνδέσουμε. Αυτό που όμως ζητούμε και επιδιώκουμε είναι επαρκής εγγύησης έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε επέθυνα και με ασφάλεια μια απόφαση καταλληλότητας. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε από τους συνομιλητές μας να μας προσφέρουν τον πιο ασφαλή και ε, δεσμευτικό τρόπο ανάληψη αυτών των ε, δεσμεύσεων. Ε, και είπατε ότι η αναλογή επιστολών δεν είναι αρκετή. Όμως υπάρχει μια ολόκληρη πυραμίδα. Η Κομισιόν καταρχήν καθορίζει τις απαιτήσει ε, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσουν οι Αμερικανικές αρχές μέσω επιστολών υπογεγραμμένων από τον αντίστοιχα υψηλότερα ιστάμενο στην ιεραρχία τους. Αυτές οι επιστολές θα εκλειφθούν ε, από τη δική μας πλευρά ως νομικά δεσμευτικές. Αναφερθήκατε στι εκλογέ. που θα λάβουν χώρα του χρόνου στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ε, ε, θα πρέπει να βασιστούμε στην συνέχεια του κράτους. Ε, γιατί αλλιώς θα πρέπει να αναστείλουμε την συμφωνία. Αυτή τη στιγμή συνομιλούμε με τη σημερινή κυβέρνηση και κάνουμε αυτό που πρέπει πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό. Ζητούμε την υψηλότερη δυνατή ιεραρχικά υπογραφή επί των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Μετά η δομή συμπληρώνεται από την απόφαση καταλληλότητας. Και σας επαναλαμβάνω, θα είναι μια μονομερής απόφαση, την οποία θα λάβει η Κομισιόν μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, η οποία θα ακολουθηθεί αν εγκρίνει την, ε, αν υιοθετεί την απόφαση η, το Κολέγιο των Επιτρόπων. Πρόκειται για μια ε, από τις πιο σοβαρές αποφάσεις που θα προτείνω, γιατί η λήψη μιας τέτοιας απόφασης θα σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε ένα τμήμα της ευθύνη για το τι θα συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όμως, χρειάζεται να λυθεί μια τέτοια απόφαση που θα βασιστεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη βέβαια η οποία θα επιβεβαιώνεται με συνεχείς ελέγχους. Η κυρία Σίπελ ρώτησε αν η, η αρμοδιότητα θα είναι σε επίπεδο κρατηδίου, ε, πολιτείας δηλαδή των πολιτιών, ή σε επίπεδο ομοσπονδιακού κράτους. Ε, αν θα είναι ένας ο διαμεσολαβητής ή ένας ανα ε, πολιτεία. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι ένας στο, σε όλη τη χώρα. Σε ό,τι αφορά την, ε, τον νόμο περί ατομικής προσφυγής, νομίζουμε ότι ο νόμος θα υιοθετηθεί σύντομα. Όλα αυτά βέβαια πλέον εξαρτώνται από την υπογραφή της συμφωνίας ε, ε, είναι ένα σχετικό, μια δύσκολη κατάσταση γιατί εμείς εξαρτάμε τη συμφωνία από το νομοσχέδιο, από τη ψήφιση του νομοσχεδίου και οι Αμερικανοί εξαρτούν τη ψήφιση του νομοσχεδίου από την υπογραφή της συμφωνίας. Ρωτήσατε επίσης ποιους αφορά αυτή η συμφωνία, ποιους καλύπτει. Ε, δεν καλύπτει μόνο τους Ευρωπαίους, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτει και όλους τους αλλοδαπούς από τρίτες χώρες. Γνωρίζω την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και θα απαντήσουμε γιατί πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς, νομίζω ότι ήδη απάντησα. Θα επιδιώξουμε ε, μια πολύ λεπτομερή και ακριβή ε, διατύπωση των περιορισμών και επαναλαμβάνω ότι μόνο η πραγματικότητα θα δείξει πώς λειτουργεί το σύστημα και θα παρακολουθούμε πολύ στενά την πραγματικότητα. Αν δούμε ότι το νέο σύστημα ε, αποτυγχάνει, θα υπάρχει συμφωνία, μια ρήτρα αναστολής που θα αναφέρει πως υπό συγκεκριμένε συνθήκες που δεν λειτουργεί το σύστημα όταν οι δεσμεύσει ε, πλευρά των ΗΠΑ δεν τηρούνται θα ανασταλεί η συνολική διευθέτηση. Ζητήσατε μια καλύτερη περιγραφή της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις αγωγές. η, το πρώτο επίπεδο λύσης είναι οι καταγγέλλοντες, οι πολίτες να απευθύνονται στις εταιρείε. Βάσει της ε, μέχρι τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των καταγγελιών αυτών επιλύονται σε επίπεδο επιχείρησης. Μετά θα υπάρχουν άλλοι τρόποι σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποτύχει. η εμπλοκή των αρχών επίλυση διαφορών, θα υπάρχουν εναλλακτικέ μορφές επίλυσης διαφορών, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η FTC. Κάποιοι ρωτήσετε ποιες αρμοδιότητες έχει αυτή η Επιτροπή. Εμείς προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την διακριτική, την διακριτική ικανότητα της ε, FTC. Αν ωστόσο η FTC δεν αντιμετωπίζει δεν εξετάσει την καταγγελία αυτή, υπάρχει ένα διαιτητικό πάνελ ως ε, ίστατος κριτής. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί περαιτέρω. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες ε, ακόμα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Ο πρόεδρος ε, ζητά λίγα λεπτά ακόμα από τη, τους διερμηνείς. Κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις, δεν ξέρω από την κυρία Έγκλεμβέλτ, ε, τι θέλει. σαν να το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είχαμε αντίστοιχε συζητήσει παλιά όταν μιλούσαμε για τη συμφωνία PNR με τη ΣΥΠΑ. Έλεγαν οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι θα αναλάβουν δεσμεύσει, δηλαδή γραπτές διαβεβαιώσει στην ουσία, που είχαμε πει ότι τότε ότι δεν είναι αρκετό και το απέρριψε το δικαστήριο. Ας μην δημιουργούμε δηλαδή νέα προβλήματα ξανά. Θέλουμε να έχουμε μία εικόνα των, ε, νομι, του νομι, της νομικής κατάστασης. Άλλο το undertaking, η ανάληψη υποχρεώσεως και άλλο οι γραπτές διαβεβαιώσεις. Ευχαριστώ πρώτα και ευχαριστώ τις Γερμηνείς. Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε να μας μιλήσετε για τις συνέπειες της απόφασης ΧΕΜΠΦ γιατί καταδίκασε η απόφαση αυτή την ε, θέση της Επιτροπής. Το λιγότερο λοιπόν θα ήταν να να δικαιολογηθείτε. Ήρθατε καθυσυχαστικοί, Εγώ ωστόσο ανησυχώ από αυτά που ακούω. Και την πρώτη φορά η καταδίκη της Επιτροπής οφείλεται στο ότι είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις και το σύστημα των ΗΠΑ. Το μόνο που πετύχατε τώρα καινούριο είναι μια ανταλλαγή επιστολών. Φλου. Μα λέτε ότι αυτό είναι καλό ο δρόμο, όλα ωραία και καλά. Δεν συμφωνώ, Επίτροπε. Νομίζουμε ότι έχουμε μπροστά μα ένα κράτο που είναι βεβαίω εταίρο, αλλά από την άλλη είχε μαζί, έκανε μαζικέ παρακολουθήσει και θα συνεχίσει να το κάνει. Όσο δεν υπάρχει αμερικανική νομοθεσία κατά τη δυνατότητα αυτή, δεν είμαι ήσυχο. Σα διαβεβαιώ ωστόσο ότι είχα πάει και προσωπικά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όπου στα πλαίσια μια κοινοβουλευτική αποστολή είδα Αμερικανού υπαλλήλου, μίλησα μαζί του για την απόφαση και τι συνέπειε που ήθελαν, τι επιπτώσει. Δεν μίλησα με τον Ομπάμπα, αλλά μπορώ να σα πω ότι δεν, είχαν, δεν πνεύμα συνεργασία. Μίλησαν για την Αμερικανική κυριαρχία και εν τέλει αυτό που μου είπαν είναι πίεση δεν δέχονται. Αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητα επίτροπε. Μήπως θυσιάζετε, επίτροπε, την προστασία μας στη βούληση να υπογράψετε την ε, συμφωνία TTIB. Αν θέλετε να κλείσετε, κλείστε. Και ευχαριστώ για τις γερμηνίες. Πού θα κάτσουν κι άλλο. Λοιπόν, τι θα πεις Βέρα. Ναι, για να απαντήσω σε αυτό το τελευταίο ερώτημα. Όχι, όχι καθόλου. Δεν θυσιάζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο βωμό αυτό. Και επαναλαμβάνω, βασικός μου στόχος και βασικός μας στόχος είναι να εγγυηθούμε αντίστοιχου επίπεδου προστασία στην Αμερικανική επικράτεια. Επειδή δεν έχουμε δικαιοδοσία λοιπόν το αμερικανικό έδαφος θα πρέπει αναγκαστικά να στηριχθούμε στις αμερικανικές αρχές να μας δώσουν τις απαραίτητες εγγύησεις και τις δικλείδες ασφαλείας. Πολύ λυπάμαι αν σας έδωσα την εντύπωση ότι οι συνομιλίες ήταν εύκολες. Καθόλου εύκολες δεν ήταν. Ήταν πραγματικά σκληρές οι διαπραγματεύσεις αυτές και εξακολουθούν να είναι έτσι. Οι συνομιλίες λοιπόν αυτές ήταν πραγματικά ε, δύσκολες, αλλά θα πρέπει να επιδείξουμε κάποιες, ε, κάποια σημάδια εμπιστοσύνη και να θέσουμε φυσικά και κάποιους κανόνες. Κανόνες οι οποίοι θα εγγυώνται τις μεγαλύτερες δυνατές εγγυήσεις για να ελέγξουμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί και εγγυήσεις για το ότι θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Επαναλαμβάνω, αν αυτό στην πράξη δεν λειτουργήσει, αυτό θα φανεί μετά από κάποιο χρόνο λειτουργία ε, τη ε, ρύθμιση αυτής. Είμαι έτοιμη να προτείνω αναστολή του συστήματος αυτού, γιατί το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι στεναρό. Δεν θα πρέπει να αποτελεί παγίδα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. <coughs> Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος, είναι εξαιρετική η κατάσταση αυτή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητάει με τα πράγματα αυτά με τους Αμερικανούς ομολόγους, αλλά δεν έχουμε ακόμα τίποτα γραπτό. Αύριο θα έχουμε ένα κείμενο. Ως πολιτικό σώμα θέλουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία αυτή σε όλα όσα συζητιούνται. Υπάρχει νομίζω ευρία συνέντευξη γι' αυτό, ότι θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασία. Αυτό ενισχύει και τις δικές σα θέσει θέσεις. Ιδιαίτερα τις προτάσεις που μας ε, αρέσουν. Γι' αυτό ζητήσαμε αναστολή το 2014 και αυτά θέλει να συζητήσει λοιπόν το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι για την ε, παρουσίασή σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και σας συναδέλφους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για το ότι αντέξετε μας τελευταία τόσο.